Καλησπέρα σα, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν θέλω να συζητήσω την κατανόησή σα γιατί είναι η τελευταία φορά που αναλαμβάνω την Προεδρία κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορίας. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στον κύριο εισηγητή, στον κύριο Φόξ. Εδώ είναι, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Uh, thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεδομένου ότι έχουμε καθυστερήσει κάπω τις διαδικασίες, θα είμαι γρήγορο να ευχαριστήσω του κοιόδη εισηγητέ, τη γραμματεία και το προσωπικό για τη συνεργασία του στην επεξεργασία αυτή τη γνωμοδότηση, καθώ είχαμε ε, και πολύ στενέ προθεσμίε για τι καλοκαιρινέ διακοπέ. Καταρχήν θέλω να αναφερθώ στη διατύπωση τη γνωμοδότηση ε, πριν να στραφούμε στα αριθμητικά στοιχεία. Γιατί αν δούμε τη διατύπωση τη γνωμοδότηση, Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε κατορθώσει να πετύχουμε ευρύ συμβιβασμού. Λέμε ότι θα έχουμε μία ε, μια προσέγγιση υπεύθυνη και θέλουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή Προπολογισμών και ε, θέλουμε να λέμε ότι έχουμε επαρκή χρηματοδότηση για το ΕΣΤΙΣ και θα ε, ταιριάξουμε αυτές τις θετικέ προοπτικές με αυτές τις αρνητικές προτεραιότητες όπως αποκαλούν κάποια μέλη, ενώ εγώ τις αποκαλώ περικοπές. Όποιο και ο και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε, είναι σαφέ ότι θέλουμε να μετακινήσουμε τις δαπάνες από ένα τομέα σε άλλον. Αλλά σε σχέση με τη διατύπωση της γνωμοδότησης, ενώ αυτή η διατύπωση είναι καλή, η όρη είναι καλή, φοβάμαι ότι κάποιες από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί δεν είναι τόσο καλές. Εγώ συμφωνώ με τις τροπολογίες για πρόσθετη χρηματοδότηση για το ΙΣΙΣ, γιατί αυτό θέτει συνάδει με την προτεραιότητα που έχουμε θέσει, αλλά αυτό που βλέπουν κάποιοι βουλευτέ σε αυτήν την Επιτροπή είναι ότι ε, κάποιοι συμφωνούν στα λόγια, ενώ όταν πρόκειται για τροπολογίες ε, ουσιαστικά ε, προτείνουν αύξηση στις δαπάνες σχεδόν στα πάντα και στρέφουμε κυρίως στις ομάδες των συλλεστών και στο ΕΛΚ και θέλω να ζητήσω κυρίως από τον κύριο Λοβίνσκεν όταν θα πάρει το λόγο να μας εξηγήσει γιατί η τροπολογία 67-20 και 67-24 είναι προτεραιότητες. Προτείνεται 2,4 επιπλέον εκατομμύρια ευρώ για ε, να απασχοληθεί προσωπικό για τις στατιστικές και στην 6724 1,7 εκατομμύρια ευρώ δαπάνες ε, σχετικά με ε, την ενεργητική απασχόληση και τα τελωνία επιπλέον προσωπικό εκεί. Όμως αυτό δεν αποτελεί η προτεραιότητα που έχουμε εμείς θέσει σε οποιαδήποτε από τις συζητήσεις μας ούτε σε κάποια γραπτή γνωμοδότηση. Και θέλω να παροτρύνω τους συναδελφούς να καταψηφίσουν αυτές τις δύο τροπολογίες. με που ο κύριος Γκοζές από το ΕΛΚ ε, υποστηρίζει αυτές τις αυξήσεις των δαπανών, γιατί σε όλες μας τις συζητήσεις είπαμε ότι θέλουμε να θέσουμε προτεραιότητες. Και αν ε, πρόκειται να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο ότι θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητες στο τότε πρέπει να το κάνουμε. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι ότι να λέμε αφενός ότι αυτή είναι η προ διάθεσή μας και κατόπιν να υπερψηφίζουμε οποιαδήποτε πρόταση εμφανίζεται για αυξήσεις. Δαπανών. Ε, ευχαριστώ τον αδελφό Γκρίνγκολτ ε, από την ομάδα των Περσιβνών για την τροπολογία που κατέθεσε που προβλέπει μείωση δαπανών 4 εκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα PRINCE ε, για την επικοινωνία για την Οικονομική και Ένωση. Θέλω οι συναδέλφοι να υποστηρίξουν γιατί, αυτή την τροπολογία, γιατί θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε 4 εκατομμύρια ευρώ εδώ και θα μπορούσαμε να τα στο ίσως. Έτσι λοιπόν ε, θα μπορούσαμε απόψε να έχουμε τελικά μία γνωμοδότηση που λέει τα σωστά λόγια, αλλά όταν φτάσουμε στα πραγματικά νούμερα, οι συνάδελφοι εδώ θα διστάζουν να ψηφίσουν οποιασδήποτε περικοπές. Και φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο μας δείχνει κάνει ανόητους. Θα ζητήσω λοιπόν από τους συναδελφούς ε, να υποστηρίξουν την 6729 ε, από τους Πρασίνων και τη δική μου 6703 και 6704 δικές μου για συγκεκριμένες περικοπές και θα τους ζητήσω να καταψηφίσουν την 6720 και την 6724 από τον κύριο Λέβιξον εκτός ε, και αν μπορεί να μας παρουσιάσει πιστικά επιχειρήματα σε σχέση με το γιατί θα πρέπει να δαπανίσουμε περισσότερα για την... Ε, ε, για, περαιτέρω προσωπικό στον τομέα της φορολογίας. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Φόξ, στη συνέχεια. Θα δώσουμε το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Θα σας παρακαλούσα να είστε όσο το δυνατόν συντομότεροι, γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε καθυστερήσει μισή ώρα ήδη. Λόγω της παρουσίασης ε, του κυρίου Μπαρνιέ. Ήταν ιδιαίτερα πυκνή. Έτσι λοιπόν, στο μέτρο του δυνατού, θα σας παρακαλούσα να είστε στο δυνατόν πιο σύντομοι. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκοζές. Παρακαλώ, Ζαν Πολύ σύντομος θα είμαι, Πρόεδρε. Να σα πω ότι ενίοτε ε, είναι πιο ενδιαφέρον να θέλουμε να ακούμε τον Επίτροπο όταν θέλει να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις ε, παρά να κοιτάμε το ρολόι και δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Και εγώ δεν ε, παίρνω το λόγο όταν μας λέτε να εκφραστούμε μόνο για 10 δευτερόλεπτα. Θα ψηφίσουμε στη συνέχεια και όπως και να έχει αυτό το εγχείρημα ουσιαστικά δεν έχει νόημα γιατί δεν θα ληφθούν καθόλου υπόψη οι δικές μας ε, απόψεις ε, και θέλουμε να μειώσουμε τις δαπάνες ε, για τους οργανισμούς ελέγχου. Έτσι λοιπόν όταν μιλάμε για την επόμενη υποπτία και για το ρόλο της EBA και όταν λέμε ότι πρέπει να μειωθούν τα νούμερα τότε εγώ αναρωτιέμαι όταν ακούω όλα αυτά ποιος λέει την αλήθεια. Ευχαριστώ κύριε Γκοζές από την ομάδα των Σοσιαλιστών, ο κύριος Λούντιξον. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή για την επικοδομητική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά είναι θετικά και χαίρομαι γιατί υπάρχει ευρεία συμφωνία στην Επιτροπή για, τις την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή που θα πρέπει να ε, με περισσότερα και όχι λιγότερα κονδύλια. Επίσης, ε, είναι σαφές ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειάζεται ισχυρότερη εποπτεία και αυτή θα πρέπει να την ε, δρομολογήσουμε με σταθερότητα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς και αλλού. Οι βασικές προτεραιότητες είναι σαφές, αλλά δεν πρέπει μέσω, λόγω αυτό να ξεχνάμε άλλους σημαντικούς τομείς. Εγώ έχω προβλέψει τρεις προτεραιότητες, δύο τις ανέφερε ο εισηγητής. Μπορούμε να κάνουμε την προσθήκη. Να διασφαλίσουμε καταρχήν ότι η Κομισιόν θα βρει τους απαραίτητους πόρους ούτως ώστε να είναι αποτελεσματική η οικονομική, ε, ο οικονομικός σχεδιασμός και η οικονομική πολιτική. Ε, υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το σχεδιασμό, συντονισμό, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Σημαντική ε, δουλειά αυτή που θα πρέπει βέβαια να ε, στηρίζεται σε ε, κατάλληλο προσωπικό και επαρκές προσωπικό. Θα πρέπει επίσης οι στατιστικές πανευρωπαϊκά να βελτιωθούν, κυρίως εις ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία, γιατί αυτό θα ε, βοηθήσει να υλοποιηθούν και άλλα προγράμματα με βάση τα μακροπρόθεσμα προγράμματα. Δεν πρέπει να μειώσουμε τη φιλοδοξία μας ούτε τους πόρους που διαθέτουμε για τα προγράμματα. Και τέλος είναι σημαντικό να καταπολεμηθεί η ε, φοροδιαφυγή. Η Κομισιόν ε, ήταν πολύ θετική στα μέτρα αυτά ενίσχυσης της πάταξης της φοροδιαφυγής θα πρέπει να βελτιώσουμε τα μέτρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα ε, δυσμενή αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται στον προϋπολογισμό μας. Ε, ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Όλες οι δαπάνες που δεν ε, δικαιολογούνται θα πρέπει να περικοπούν βέβαια δεν θα πρέπει να κάνουμε περικοπές σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού και να ζημιώσουμε έτσι ε, το στόχο μας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τόνωση της οικονομίας. Αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό. Προσοχή λοιπόν, δεν πρέπει να κάνουμε μειώσεις και περικοπές που θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο. Αυτά. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια από τους φιλελεύθερους, ο κύριος και πάλι θα σας παρακαλούσα να είστε πάρα πολύ σύντομος, γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, έτρεχα για να προλάβω και λαχάνιασα. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Είναι πάρα πολύ ε, ισορροπημένη η γνωμοδότηση. Για τα νούμερα συμφωνούμε όλοι ότι η οικονομική αρχή επιτήρησης ε, θα πρέπει να προχωρήσει πέρα από τις προτάσεις της Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τον λοιπό προϋπολογισμό, όπως ε, υπάρχει στο κείμενο της γνωμοδότησης, ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύ, τις πολύ καλά διατυπωμένες συμβιβαστικές λύσεις που αντικατοπτρίζουν τις απόψεις όλων μας. Χρειάζεται υπεύθυνο προπολογισμό με σαφεί προτεραιότητε, Πρέπει να έχουμε θάρρος να περικόψουμε γραμμές λιγότερο σημαντικές και θα πρέπει να ε, εκπληρώσουμε τους ε, στόχους της στρατηγικής 2020. Όμως, ε, αν και βλέπω το πολιτικό όφελος της πρότασης, θα ήμουν κατά του οριζόντιου παγώματος του προϋπολογισμού γιατί το, οι τωρινέ ανάγκες πληρωμών ε, έχουν συμφωνηθεί και έχουμε συμφωνήσει δυο φορές πάνω σε αυτές και στο προηγούμενο ε, ετήσιο προϋπολογισμό. Πρέπει λοιπόν τώρα να τα υπομισθούμε αυτά. Επίσης δεν συμφωνώ απόλυτα να αυξηθεί ο, ο προϋπολογισμός της Ένωσης ε, όπως αναφέρθηκε στην ε, περσινή έκθεση ε, για την κρίση. Η προτινόμενη αύξηση δεν είναι σόφρον και είμαι κατά της ε, σχετικής τροπολογίας. Δεν θέλω να συμπεριληφθεί στη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Αυτά είχα μόνο να σας πω. Ευχαριστώ κύριε Τόρβαλτς. Κύριος Διχόλ. Κοιτάξτε. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για τη συνεργασία που είχαμε ή που ακούω ότι υπήρξε. Συμφωνήσαμε σχεδόν σε όλα, στα κυριότερα τουλάχιστον και οι συμβιβαστικές τροπολογίες το δείχνουν. Η μόνη διαφωνία αφορά τη συμβιβαστική α που λέει βασικά ότι όλες οι αυξήσεις πρέπει να αντιστοιχούν σε περικοπές. Αυτό αντιφάσκει με γνωστή θέση του Κοινοβουλίου που έλεγε ότι και για μακροοικονομικούς λόγους και για άλλους η εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς πρέπει όλο και μεγαλύτερο ευρωπαϊκό, υψηλότερο ευρωπαϊκό προπολογισμό βήμα με το βήμα. Και αυτό δεν είναι κάτι πολύ πολύ πολύπλοκο. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε θρησκευτικά αυτά τα πράγματα. Υπάρχει η Σιλβί Κουλάρ, οι σοσιαλιστές και από τη δική μας ομάδα προτάσεις να πάψει πια να ισχύει αυτό το δόγμα ότι ο ευρωπαϊκός προβλογισμός δεν μπορεί και δεν πρέπει να αυξηθεί και ότι κάθε αύξηση πρέπει να αντιστοιχεί σε περικοπή. Παρακαλώ λοιπόν τους συναδέλφους εδώ να αλλάξουν τη θέση τους για το συμβιβασμό α, για τη συμβιβαστική α, γιατί αντιφάσκει με παλιότερα μας ψηφίσματα αφού θέλουμε όλο και ισχυρότερη κοινή αγορά. Από την ΚΟΕ δεν βλέπω τον κύριο Κλούτε. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Σαμποτέρο από το EFD. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Φόξ για την εξαιρετική δουλειά του ως εισηγητή. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, εγώ θεωρώ ότι είναι σοφρόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει το καλό παράδειγμα. Έχουμε αυστηρά μετρελαιτότητα στα κράτη-μέλη, γι' αυτό υποστηρίζω την άποψη του εισηγητή, ο προπολογισμός του 2013 να παγώσει Όμω, με ανησυχούν ορισμένε τροπολογίε που έχουν κατατεθεί και που αντιτίθενται στην αρχή αυτή και ίσως να αναγκαστώ να καταψηφίσω την έκθεση αυτή ακόμη και αν ε, προετοιμάστηκε τόσο καλά. Στο μέλλον, ε, όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θυμούνται ότι δεν είναι ατελειωτοί πόροι και όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις πάντοτε θα υπάρχει και κόστος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φόξ, θέλετε να επανέλθετε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι θα ήθελαν να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στην ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε καταρχήν τη γνωμοδότηση, αλλά να δούμε καταρχήν να κάνουμε μια δοκιμή με τις κάρτες σας, αν μπορείτε. Να βάλετε τις κάρτες, να τοποθετήσετε τις κάρτες σας για να κάνουμε μια δοκιμή. Todavía faltan seis personas. Λείπουν έξι άτομα. Okay. It's okay. Εντάξει είναι. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στη ψηφοφορία της ε, γνωμοδότησης, στην τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είστε προηγούμενος έλεγχος. Πέρας της ψηφοφορίας. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Να προχωρήσουμε στην τροπολογία 2. 3. Υπέρ. Όχι, 2 διορθώνει ο Πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά αποχές για να ελέγξουμε. We close. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Εποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για να ελέγξουμε. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Yeah, okay, so this doesn't change. Και εγώ ψηφίζω, λοιπόν πρέπει να το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη. Συμβιβασμός Α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10, συγγνώμη. Συμβασμός Α, λέει ο Πρόεδρος. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμούς Β. Υπέρ. Εδώ Έχουμε μια τμηματική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεσμός Γ, Σ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπο... Συμβιβασμός D, δέλτα, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Συνδεσμός Ή, ε, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 38. 39. Συγγνώμη, 39. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Την 39 ψηφίζουμε.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 37 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές. Ας προχωρήσουμε στο επιλογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κοινωνικό έτος 2013. Υπολογία 6726 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6729 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εκδόθησαν ή δεν μηδέν; Είμαι κάποιος κατά της πρότασης αυτής. So we go now to 01. Να περάσουμε στην 6701, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 6719, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Για να ελέγξουμε την 6719. Αρχή τη ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Agreed. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Ψηφίσαμε την 67.001. Ναι. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί. Αφού απορρίφθηκε η δική μου τροπολογία, νομίζω ότι έπρεπε να ψηφιστεί. Απορρίφθηκε. Ψηφίσαμε και απορρίφθηκε η δική μου απερίφθη, αλλά όχι αυτή του συγητή νομίζω. Να την ξαναδούμε, υπέρ. Για την 67.00, για να αποσαφηνίσουμε. Κατά, εποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε, συγγνώμη. πέρας τη ψηφορία. Those in favor. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Συγγνώμη. Καταπίπτει. 0-2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Συγγνώμη. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64-41 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Είπα ότι υιοθετήθηκε, αλλά να το δούμε. We open the votes, we close. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Άρα cual... Amendment number 40. Τροπολογία 42, υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 03 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 04 υπέρ κατά αποχές 7000. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 05 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη για τα λάθη μου και περνάμε στο επόμενο σημείο.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 να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Στο επόμενο σημείο ζητώ συγγνώμη από τον Επίτροπο Λένε για την καθυστέρηση που σημειώθηκε απόψε και χωρίς χρονοτριβή θα δώσω το λόγο στον κύριο Επίτροπο για να μας παρουσιάσει πώς ε, βλέπει τη μελλοντική οικονομική και νομισματική ένωση. Παρακαλώ έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι άρχισε με πολύ ε, βαρύ και πολύ άσχολο τρόπο αυτή η σεζόν Ευχαριστώ για την ε, πρωτοβουλία, για τη συζήτηση αυτή, για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, που είναι ένα εγχείρημα ε, ε, επί του οποίου εργαστήκαμε από κοινού τα προηγούμενα δυόμιση χρόνια και το οποίο θα συνεχίσουμε να το επεξεργαζόμεθα τουλάχιστον για τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Πιστεύω ότι μια ενδελεχή συζήτηση για αυτά τα θέματα είναι σημαντική ε, στα πλαίσια ενός φθινοπόρου φορτωμένου με δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια προχώρησε σε ουσιαστικά και ευρύτατα μέτρα για να καταπολεμήσει την ε, ε, κρίση του χρέους και την χρηματοπιστωτική κρίση και να βελτιώσει τη διακυβέρνηση στην Ένωση. Όμως ε, έχουν ενταθεί τον ε, προηγούμενο χρόνο τα προβλήματα, οι οικονομικές ανισορροπίες επιμένουν και αυτό σημαίνει ότι και η Νομισματική Ένωση και το μέλλον των πολιτών μας θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται υπό σοβαρές πιέσεις. Σίγουρα χρειάζονται αλλαγές στην τωρινή μας αρχιτεκτονική για να αντιμετωπίσουμε τα ε, υπόλοιπα αδύναμα σημεία στην ε, ε Οικονομική και Νομισματική Ένωση και να ενισχύσουμε ε, τα θεμέλια και να τα κάνουμε πιο στέρεα, ούτως ώστε να είναι βιώσιμη η Ευρώπη και το κοινό νόμισμα. Χρειάζεται βραχυπρόθεσμη δράση για να ανασχεθεί η κρίση, να αναζωογονηθεί η ανάπτυξη και να εξαλειφθούν οι ανισορροπίες. Και αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με μακροπρόθεσμο όραμα για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση και με σαφή οδικό χάρτη. Πάνω σε αυτή τη βάση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε ανταλλαγή απόψεων για την περαιτέρω εμβάθυνση της, Ευρωπαϊ... Ε, και Νομισματικής Ένωσης, της ε, ΟΝΕ. Ο πρόεδρος Φαν Ρομπάι το παρουσίασε σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Eurogroup και της ε, Κεντρικής Τράπεζας. Τέσσερα είναι τα βασικά δομικά στοιχεία για το μέλλον τη ΟΝΕ. Ε, ένα ολοκληρωμένο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, ένα ε, ολοκληρωμένο πλαίσιο προϋπολογισμού, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής και βελτιωμένη λογοδοσία και δημοκρατική νομιμοποίηση. Χρειάζονται πρόοδοι σε όλα αυτά τα θέματα και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έδωσαν μια εντολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μαζί με τους τρεις προέδρους ε, να παρουσιάσει μια ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης τον Οκτώβριο και μια τελική έκθεση πριν από το τέλος αυτού του έτους. Η ενδιάμεση αξιολόγηση, έκθεση, θα επικεντρώνεται σε περαιτέρω μέτρα που μπορεί να ληφθούν βράχη πρόθεσμα ενώ η τελική έκθεση το Δεκέμβριο θα εξετάζει και το τι μπορεί να γίνει στο πλαίσιο, το υφιστάμενο πλαίσιο της συνθήκης και ποια μέτρα θα απαιτήσουν αλλαγές στη συνθήκη. Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προφανώς θα ενέχονται στενά στις διαδικασίες αυτές, στην προβληματική αυτή και θα γίνονται διαβουλεύσεις κατά την προετοιμασία των εκθέσεων. Ο στόχος της διαδικασίας διαβουλεύσεων είναι να δημιουργηθεί συνένεση όπου είναι αυτό εφικτό βραχυπρόθεσμα και όπου είναι αυτό επιθυμητό πιο μακροπρόθεσμα, ούτω ώστε να καταλήξουμε σε ένα συνεκτικό δικό χάρτη για την επίτευξη γνήσιας Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ειδικά αυτό σημαίνει την ολοκλήρωση της αναδόμησης της ΟΝΕ που λαμβάνει η χώρα τώρα για να δημιουργηθεί ε, μια νέα ΟΝΕ πολύ διαφορετική από αυτή που είδαμε την πρώτη δεκαετία της ύπαρξης της ΩΝΕ. Αξιότιμα κράτη-μέλη, η περαιτέρω ε, ανάπτυξη της ε, ενοποίησης των τραπεζών, της, δημοσιο... της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, είναι πολύ σημαντική στην προσπάθειά μας. Πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς καθυστέρηση σε δύο στάδια. Τώρα είμαστε στο πρώτο στάδιο Παράλληλα με τη δήλωση από τις 29 Ιουνίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Κομισιόν εργάστηκε πάνω σε μια νομοθετική πρόταση για την δημιουργία ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού για τις τράπεζες της Ευρωζώνης. Αυτό θεωρείται θέμα κατεπήγων. Θα παρουσιαστεί το θέμα σε λιγότερο διάστημα των δύο εβδομάδων, ε, μέσα σε δέκα μέρες ε, συγκεκριμένα, για να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, να οριστικοποιηθεί. Συμφωνία για ενιαίο εποπτικό μηχανισμό θα ε, ετοιμάσει το έδαφος για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, τον ESM, ούτως ώστε να έχουμε ένα νέο μέσο που, και, να έχουμε ένα νέο μέσο που θα επιτρέπει την άμεση ανακεφαλαιοποίηση, την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ε, αν η, περάσει η υποπτία των τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν προχωρήσουμε ε, στα βήματα που χρειάζονται για να έχουμε μια πλήρη τραπεζική ένωση, ενοποίηση, αυτά είναι σημαντικά για τη σταθερότητα της ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής οικονομίας και να σπάσουμε αυτόν τον αρνητικό, το φαύλο κύκλο αυτό μεταξύ ε, δημοσίου, κυβερνήσεων και τραπεζών που βλάπτει την ευρωπαϊκή οικονομία και την δυνατότητα που έχει να αυξάνεται, να αναπτύσσεται και να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Ξέρω ότι συζητήσατε τα επιμέρους αυτού του θέματος με τον συνάδελφο Μπαρνιέ και είναι και θέμα βέβαια ε, που απασχολεί και τον πρόεδρο Μάριο Ντράγκη. Και με τους δύο έχω συνεργαστεί στενά. Αν αυτό θέλετε να το θεωρήσετε ως ένδειξη ενότητας και αμοιβαίας κατανόησης, δεν με πειράζει. Θα ήθελα να παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία της πρότασής μας επειδή είναι ακρογωνιαίος λίθος αυτός, αν όχι ο ακρογωνιαίος λίθος στην συνολική μας αντίδραση στην κρίση και το μέλλον της, Ευρωπαϊ... της ΟΝΕ ναι και του Ευρώ. Το σημείο εκκινήσεως είναι ότι ε, θα πρέπει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι υψηλή ολοκλήρωσης παρόλο που είδαμε και σαφή δείγματα ε, πανεθνικοποίησης ε, τον τελευταίο χρόνο λόγω της κρίσης. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μεγάλη, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες, υπάρχει ε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η χρηματοπιστωτική αστάθεια να ε, μολύνει άλλες χώρες από μια χώρα. Ε, η διασυνοριακή αυτή μετάδοση της κρίσης είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν μιλάμε για τις χώρες της Ευρωζώνης. Ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός θα ισχύει λοιπόν ε, για όλα τα κράτη της Ευρωζώνης, αλλά θα είμαστε ανοιχτοί για τη συμμετοχή και άλλων κρατών που θα θελήσουν να ακολουθήσουν αυτή την πορεία της βαθύτερης ολοκλήρωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να αναλάβει μια νομική δέσμευση και να δώσει διασφαλίσεις ότι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αυτά τα πλαίσια θα είναι δεσμευτικές για τις εθνικές αρχές και τις τράπεζες. Ο ενίος εποπτικός μηχανισμός θα πρέπει να έχει φιλόδοξο πρόγραμμα εις ό,τι αφορά τον αριθμό των τραπεζών που θα καλύπτει. Όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια, ακόμα και μικρές ή μεσαίες τράπεζες μπορεί να είναι συστημική σημασίας και μπορεί να δημιουργήσουν κοινωνικές αναταραχές και προβλήματα. Μιλάω για την Northern Rock, την ε, Anglo-Irish ή την Bankia. Η προσέγγιση μας λοιπόν προβλέπει έναν φιλόδοξο μηχανισμό με ευρεία κάλυψη που θα καλύψει όλες τις τράπεζες στην Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι στην καρδιά του όλου συστήματος. Η ΕΚΤ λοιπόν θα πρέπει να έχει την πρωταρχική ευθύνη και βασικά κέρια καθήκοντα εποπτείας για αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας εποπτεία οι εθνικές εποπτικές αρχές που έχουν αποκτήσει πείρα και έχουν αναπτύξει πραγματογνωμοσύνη ε, στην ε, προληπτική εποπτεία θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στο μελλοντικό αυτό Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τυχόν κίνδυνη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των φορέων λήψεως αποφάσεων της ΕΚΤ θα απαλληφθεί, δεν θα υφίσταται, κυρίως γιατί θα έχουμε ε, διαχωρισμό των εποπτικών αρχών από τις αρχές υπεύθυνες για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Τέλος, κατάλληλοι μηχανισμοί δημοκρατικής λογοδοσίας πρέπει να δημιουργηθούν για τα εποπτικά καθήκοντα η ευθύνη της ΕΚΤ θα πρέπει να ενισχυθεί σε σύγκριση με τη, δηλαδή θα πρέπει να ενισχυθεί η λογοδοσία της ΕΚΤ σε σύγκριση με την ανεξαρτησία της στον τομέα της νομισματικής πολιτικής. Η Κομισιόν έχει προτείνει, όπως γνωρίζετε ήδη, νομοθεσία που θα ενισχύσει τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα για τα προγράμματα ε, εγγύησης καταθέσεων και την εξυγίανση και ανάνυψη των τραπεζών και για να ε, βελτιωθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών. Όλα αυτά θα ισχύουν για τους 27 αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει τα μέτρα να εγκριθούν από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατόν. Στο δεύτερο στάδιο θα πρέπει να επιτελέσουμε αποφασιστική πρόοδο ούτως ώστε να έχουμε κοινό πρόγραμμα ε, εγγύησης των ε, καταθετών των καταθέσεων και των καταθετών για μια, ένα ενιαίο πλαίσιο εξυγένσης και ανακάμψης. Ε, παρουσιάζοντας την νομοθετική πρόταση και αυτό θα γίνει όπως είπα τις επόμενες δύο εβδομάδες ή δέκα μέρες για την ε, δημιουργία ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού θα εγκρίνουμε επίσης και μία ανακοίνωση που θα ε, σκιαγραφεί τον οδικό χάρτη προς μια ολοκληρωμένη τραπεζική ενοποίηση. Ε, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, τα πολύ υψηλά επίπεδα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής ε, αλληλεξάρτησης ε, απαιτούν ένα ποιοτικό βήμα προς την Δημοσιονομική Ένωση, ούτως ώστε να ε, λειτουργεί όσο γίνεται πιο απρόσκοπτα η ΟΝΕ προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Μία δημοσιονομική ένωση θα πρέπει να διασφαλίζει πιο χρηστή δημοσιονομική πολιτική σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτω ώστε να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και να διασφαλίζει τη μακροοικονομική σταθερότητα πρέπει να περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την πρόληψη και διόρθωση των μη βιώσιμων δημοσιονομικών εξελίξεων στα κράτη-μέλη και πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και μέσα και μηχανισμούς για να αντιμετωπίζει ασύμετρα οικονομικά σοκ και να προλαμβάνει την μετάδοση των κρίσεων και προβλημάτων στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει ε, συντονισμένη ή κοινή αλλά περιορισμένη έκδοση ομολόγων ε, και βέβαια και ο επιμερισμός του κινδύνου συνοδεύεται με ε, παράλληλα μέτρα ε, βελτίωσης του προϋπολογισμού, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε ε, κινδύνους και εκτροπές. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά δεν πρέπει να βάλουμε πολύ ψηλά τον πύχη, τουλάχιστον βράχη πρόθεσμα, γιατί αυτό θα μπορούσε να μας ρίξει στα χέρια εκείνων που ε, θεωρούν ε, αδύνατη την ε, γνήσια ε, οικονομική και νομισματική πολιτική. Ενώ λοιπόν εξετάζουμε, μελετούμε και δουλεύουμε πάνω στην καινούργια αρχιτεκτονική της ΟΝΕ, πρέπει ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε απόλυτα τα υφιστάμενα μέσα, την υφιστάμενη εργαλειοθήκη μας και το υφιστάμενο πλαίσιο που έχουμε ήδη θεσπίσει και να εργαστούμε για την βελτίωση και ουσιαστικά ε, και σε νομικό επίπεδο επίσης. Και έτσι φτάνω σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο δεν πρέπει να το ε, παραβλέψουμε. Θα πρέπει να βελτιώσουμε το πλαίσιο της διακυβέρνησης, ενώ ολοκληρώνουμε την εργασία για τη δέσμη των δύο μέτρων, το ΤΟΥΠΑΚ, και αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια της υφιστάμενης συνθήκης. Θα πρέπει να εισαγάγουμε νέο δυναμισμό στους συνεχιζόμενους τριμερείς διαλόγους, ούτως ώστε γρήγορα να καταλήξουμε σε συμφωνία, η οποία θα σέβεται τον αρχικό στόχο των προτάσεων και ουσιαστικά θα βελτιώνει την ε, επιτήρηση, την, ε, την εποπτεία του προϋπολογισμού και τον συντονισμό των πολιτικών μας στην Ευρωζώνη. Πρέπει λοιπόν έγκαιρα τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τα σχέδια προϋπολογισμού τους ε, για, για να εγκριθούν από τα κοινοβούλια και αποτελεσματικότερο πλαίσιο για να είμαστε βέβαιοι ότι θα διορθώνονται τα υπερβολικά ελλείμματα. Άλλα βήματα προς την ε, ολοκλήρωση μπορούν να γίνουν πιο μακροπρόθεσμα και αυτά περιλαμβάνουν ε, μεγαλύτερη ε, δημοσιονομική ολοκλήρωση, παράλληλα ενδεχομένως με κοινά μέσα αντιμετώπισης του χρέους, αλλά πρέπει να είναι σαφές ότι αυτά τα βήματα θα πρέπει να απαιτήσουν πρώτα πολύ σημαντική περαιτέρω συνένωση των φορέων λήψης αποφάσεων και όλα τα μέτρα για την πολιτική νομιμότητα και νομιμοποίηση των ε, προτάσεων αυτών θα πρέπει να ληφθούν. Αξιότιμα μέλη, ε, προχωρώ σε περαιτέρω αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την δημοσιονομική και οικονομική πολιτική ε, θα απαιτήσουν πιο ισχυρούς μηχανισμούς για να νομιμοποιήσουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται ε, από κοινού και να διασφαλίσουν τη δημοκρατική λογοδοσία και πολιτική συμμετοχή. Αυτό είναι σημαντικό για να υπάρξει και η υποστήριξη από την κοινή γνώμη ε, σημαντικών αποφάσεων που θα επηρεάσουν τόσο πολύ την καθημερινότητα των πολιτών μας. Ο οικονομικός διάλογος, ο οποίος άρχισε από τη δέσμη των 6 μέτρων, το Six Pack, είναι ένα νέο διοργανικό μέσον που διασφαλίζει ένα φόρουμ για δημοκρατική λογοδοσία στο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Ε, ένα μια ευρύτερη δυναμική του Six Pack είναι οι καινοτόμες διατάξεις που επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο, σε εσά δηλαδή, να διεξάγεται οικονομικό διάλογο με μεμονωμένα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα όταν αυτά παραβιάζουν τους νοσιακούς κανόνες του Συμφώνου ε, Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή όταν υπάρχουν ε, δημοσιονομικές ανισορροπίες. Αυτή η διάταξη επιτρέπει σε μια εθνική κυβέρνηση να ε, θεωρηθεί ότι πρέπει να λογοδοτήσει στο Κοινοβούλιο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Νομίζω ότι είναι σωστό να πούμε ότι ο οικονομικός διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μάλλον δεν αρκεί για να αντιμετωπίσουμε ε, ζητήματα δημοκρατικής νομιμότητας των Βρυξελών προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη και στενότερη συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτά τα πλαίσια να επιστήσω την προσοχή σας επίσης σε μια σημαντική πρόταση που υπάρχει στη δέσμη των δύο μέτρων, το ΤΟΥΠΑΚ, δηλαδή τη δυνατότητα η Κομισιόν να κληθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια να εξηγήσει τη θέση της, τη θέση της Κομισιόν επί των εθνικών προϋπολογισμών τη μελλοντική νομοθεσία για τη, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν τέτοιες ε, διατάξεις για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής στο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, πριν ε, αρχίσει μια γενική συζήτηση με σχόλια και ερωτήσεις, θα ήθελα να ολοκληρώσω με κάποιες σύντομες παρατηρήσεις γενικότερης φύσεως. Νομίζω ότι είναι θετικό και πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η σοβαρή συζήτηση για το μέλλον του ευρώ. Ε, τώρα άρχισε και χρειαζόταν πάρα πολύ. Περισσότεροι συμμετέχοντες στη συζήτηση συμφωνούν ότι η βαθύτερη ολοκλήρωση αποτελεί σημαντικό κομμάτι ε, για το στόχο αυτό δεν είναι αυτό το μόνο, αλλά είναι σημαντικό. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία στη λήψη των αποφάσεων. Ε, οι περισσότεροι συμμετέχοντες στη συζήτηση συμφωνούν για τη βαθύτερη ολοκλήρωση και την μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία. Και συμφωνώ και εγώ προφανώς με αυτούς. Πιστεύω ότι ε, προχωρώντας με το κοινό όραμά τους οι Ευρωπαίοι δεν μπορεί να διαιρούνται σε νικητές και ιτημένους είτε όλοι θα κερδίσουμε θα νικήσουμε όλοι μαζί ή θα χάσουμε όλοι μαζί αν ε, υπάρχει εντύπωση ότι κάποιοι αποκομίζουν ωφέλη σε βάρος των άλλων τότε το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι βιώσιμο πολιτικά ε, ήδη δυστυχώς βλέπουμε κάποια ανησυχητικά δείγματα τέτοιων ε, συναισθημάτων που θα τα γνωρίζετε κι εσείς βέβαια. Σε αυτά τα πλαίσια ε, θα πρέπει να πέσουν γέφυρες στην Ευρώπη για να γεφυρωθούν οι διαφορές, οι αντιτιθέμενες αντιλήψεις. Οι διαφορετικές αντιλήψεις θα πρέπει να αντικατασταθούν από κοινό όραμα προς μια γνήσια και αποτελεσματική οικονομική δημοσιονομική ένωση που θα στηρίζεται, όπως σας είπα, από μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία. Έτσι θα έχουμε μια ε, ένωση σταθερότητας και αλληλεγγύης που θα μπορεί να διασφαλίσει ε, βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, ΕΚΟΝ, μέλη του Κοινοβουλίου, η συμβολή σας στη συζήτηση και το όραμά μας θα είναι ουσιώδης και κέρια για το όφελος της Ευρώπης και των πολιτών της. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Τώρα θα ακούσουμε τους συναδέλφους. Έχουμε τη συζήτηση της έκθεσης Tyson και μετά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όπως και πριν, πρώτα οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων, μετά συντονιστές ή αλλά παρακαλώ να μου λέει ο καθένας τι είναι όταν εκφωνώ τα ονόματα, η Μαριάν πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο που δέχτηκε να προσέλθει. Είναι κάτι πολύ θετικό αυτές οι ανταλλαγές απόψεων και οι συναντήσεις. Κύριε Επίτροπε, το Κοινοβούλιο αποφάσισε με βάση το έγγραφο του κ. Βαν Ρόμπουι, όπως το ονομάσατε και μόνος σας προηγουμένως, να θεωρήσει το έγγραφο αυτό, όπως και τα άλλα όργανα, ως πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε προς τις καυτές εξελίξεις του καλοκαιριού. Η έκθεση βέβαια θα πρέπει να περάσει με πλειοψηφία στο από το Κοινοβούλιο και το καλοκαίρι που είναι όλοι στην άδεια δεν ε, είναι εύκολο να πάρουμε τη γνώμη των συναδέλφων. Μαζί με τη γραμματεία λοιπόν ε, αποφάσισα να περιοριστώ σε ένα έγγραφο εργασίας το οποίο περιέχει πάρα πολλές ερωτήσεις και μετά από τη συνεδρίαση αυτή θα αρχίσω να ε, φτιάχνω το σχέδιο της έκθεσης. Υπάρχουν πολλά θέματα, πολλές ερωτήσεις. Απαντήσεις ακόμα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά λεπτά και ευαίσθητα σημεία. Δεν θα τα παρουσιάσω όλα γιατί έχουν αναφερθεί κάποια, να μην επαναλαμβάνομαι, αλλά νομίζω ότι την ιδιαιτερότητα της κατάστασης την καταλαβαίνουν οι συνάδελφοι. Ε, εκεί θα στηριχτώ. Και ελπίζω ότι θα τύχει ευρεία πλειοψηφία η έκθεση, γιατί και ως Κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Με τον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας κάναμε μια ανταλλαγή απόψεων, το ίδιο και με τον Επίτροπο Μπαρνιέ και χαιρόμεθα που μπορούμε και μαζί σας να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή. Αυτό που διαπίστωσα ε, μέχρι τώρα κύριε Επίτροπε, είναι ότι υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες. Όχι τόσο σε σχέση με τα τέσσερα δομικά στοιχεία του πακέτου που αναφέρατε, την νομιμότητα, την νομιμοποίηση, τη δημοκρατική, τη λογοδοσία, αλλά ε, υπάρχει ένα πρώτο ερώτημα που αφορά την εποπτεία, την ενιαία εποπτεία των ε, τραπεζών στην Ευρώπη που θα πρέπει να στηρίζεται στο άρθρο 127 για να, ε, ε, και να κάνει, να ετοιμάζει γνωμοδοτή στο Κοινοβούλιο. Θα παραμείνει το 127 ή μήπως με δημιουργικό πνεύμα μπορούμε να στηρίξουμε σε άλλο άρθρο τη διαδικασία αυτή όπως έχει γίνει και σε άλλες εκθέσεις ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς να ασκήσουμε το νομοθετικό μας έργο. Ή θα... Ε, ε, ε, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Πώς μπορεί να ανταποκριθεί και να ασκήσει τα καθήκοντά του και τις αρμοδιότητες του Κοινοβούλου. Αυτό είναι μια ανησυχία που έχουμε όλοι. Τώρα για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Όταν πρόκειται για τραπεζική ενοποίηση με διαφορετικούς πυλώνες, Όπως ακούσαμε και από τον κύριο Μπαρνιέ και το είπατε και εσείς, ακούμε ότι θα υπάρχει η Ευρωζώνη και δυνατότητες opt-in, να μπουν και άλλοι που θέλουν. Ελπίζω να είναι πολλοί αυτοί που θα θελήσουν να μπουν, γιατί πρέπει να υπάρχει συνοχή. Μακάρι να είναι και 27 ε, που θα θελήσουν να, να προσχωρήσουν. Όσο γίνεται περισσότερα κράτη-μέλη που θα λειτουργούν όλα με τους ίδιους κανόνες. Και βέβαια, αν χρειάζονται ιδιαίτεροι κανόνες για να υπάρχει συνοχή στην Ευρωζώνη, θα πρέπει να ψηφιστούν οι κανόνες αυτοί. Θα υπάρχει δυνατότητα opt-in, ε, θα πρέπει να υπάρχει Ευρωζώνη συν δηλαδή, ούτω ώστε να προσθεθούν όσο γίνεται περισσότερα ε, κράτη-μέλη ακόμη για την ολοκλήρωση. Τώρα για την εποπτεία, ε, Europlus είναι μια επιλογή που αναφέρθηκε, το Europlus έτσι κατάλαβα δηλαδή σήμερα, αλλά μένα με ενδιαφέρει και η δική σας γνώμη. Χρειάζεται κάποια συμμετρία για το πεδίο εφαρμογή του ε, ψηφίσματος και για ε, τον πυλώνα γήσεις καταθέσεων και για τον πυλώνα εξυγίανσης. Ε, είναι το ίδιο πεδίο εφαρμογής όπως στην ε, εποπτεία θα είναι ευρύτερο αυτό το δεύτερο πεδίο εφαρμογής ή πιο στενό. Επίσης, η αρμοδιότητα της εποπτείας ε, υπάρχουν πάρα πολλές και διαφορετικές τράπεζες στα κράτη-μέλη. Ποιες εννοούμε, ποιες είναι οι τράπεζες αυτές που θα είναι υπό εποπτεία. Θα είναι όλες, αλλά για συγκεκριμένες μόνο εργασίες τους, γιατί τα ακούσαμε και αυτό. Ε, άλλοι είπαν ότι θα υπάρχει ένα ε, σύστημα που θα προβλέπει ε, διαφορετική κατανομή ανάλογα με την τράπεζα και κάθε τράπεζα θα κρίνεται χωριστά. Θα ήθελα την γνώμη σας, τι, τι, διαδικασία θα ακολουθηθεί για τις τράπεζες. Μια άλλη ανησυχία που έχουμε και όχι μόνο εμείς είναι η νομισματική εποπτεία της ΕΚΤ για νομισματικά θέματα. Για νομισματικά θέματα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη η ΕΚΤ. Αυτό το υποστηρίζουμε. Αλλά προκειμένου περί της εποπτείας πρέπει να υπάρχει λογοδοσία. Αυτό πώς θα το ρυθμίσουμε. Αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εσωτερική αρχιτεκτονική της ΕΚΤ και θα ήθελα και πάνω σε αυτό τη γνώμη σας. Και κάτι τώρα για τις σχέσεις μεταξύ ΕΚΤΕ και Τραπεζικής Αρχής, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και της ε, Κεντρικής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα, ως εποπτεία η ΕΚΤ, αν θέλουμε να εγγυηθούμε την, ε, την ε, ενιαία αγορά, τους κανόνες που πρέπει να είναι οι ίδιοι, κάποια στιγμή θα υπάρξει ανάγκη για διαμεσολάβηση μεταξύ της ε, τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ και άλλων που είναι εκτός ευρωζώνης, που δεν είναι μέσα στο σύστημα. Και αν χρειαστεί κάτι τέτοιο, τότε ποιος θα διαμεσολαβήσει, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και εν τη αυτή περιπτώσει ιεραρχικά θα είναι ανώτερη η Τραπεζική Αρχή από την ΕΚΤ. Θα πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί υπάρχουν πολλά επιχειρήματα που θα μπορούσε κανείς να διατυπώσει εδώ. Επίσης σημαντικό είναι ε, και κάτι ακόμα. Όταν θα έχουμε την εποπτική αρχή, αρκεί αυτή και ο ESM θα μπορέσει να αναλάβει τις νέες λειτουργίες, να έχει πρόσβαση δηλαδή σε τραπεζικά κεφάλαια ή θα πρέπει να περιμένουμε κι άλλο μέχρι ότου ολοκληρωθούν και οι άλλοι δύο πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης. Ελπίζω όχι. Ελπίζω μόλις ολοκληρωθεί η εποπτεία να μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Τώρα για την εγγύηση των καταθέσεων και την εξυγίανση. Δεν έχω ξεκαθαρίσει τι γνώμη έχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Εμείς είπαμε, είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ταμείο, θα είναι πολύ θετικό αυτό, αλλά το ταμείο αυτό, ή μάλλον δύο χρειαζόμαστε θα έλεγα. Ένα για την ε, διεκπεραίωση και ένα για την καθαυτό εγγύηση των καταθέσεων. Γιατί τότε και ο καταθέτης, ο αποταμιευτής θα νιώθει πιο ασφαλής να μην ε, ε, ε υπάρξει πρόβλημα δηλαδή ε, με τις καταθέσεις. Και γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα. Μια άλλη ερώτηση. Αν μιλάμε για Μιλάμε για τραπεζική ένωση, αλλά πολύ ευρέω. Δηλαδή, ευρωζώνη συν άλλε χώρε. Αλλά. Επομένω, ε, για ποιο μηχανισμό μιλάμε. Αναφερθήκατε σε ένα backstop, σε ένα μηχανισμό υποστήριξης. Ε, θα λειτουργεί δηλαδή ο ΣΕΜ σε μηχανισμό υποστήριξης για τις 17 ε, χώρες μόνο ή και για χώρες που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Ούτε αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρο. Σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση αυτά, σε ό,τι αφορά τώρα ε, το μας είπατε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Θα υπάρχει και ένας τριμερής διάλογος αύριο για το και Ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε τα θέματα αυτά σε πρώτη ανάγνωση για την ε, σύνοδο, αν εκφραστεί εκεί η βούληση να προχωρήσουμε, δεν ξέρω αν ε, μπορεί οι κομισιόνες της τις κυβερνήσεις να παρουσιάσουν ε, εκ των προτέρων ε, τα προγράμματα για τον προϋπολογισμό, αλλά και ακόμη και αν ψηφιστεί ο προπολογισμό από το Κοινοβούλιο, αν κάτι δεν πάει καλά, τότε θα πρέπει να μπορούμε να πούμε σε εκείνη τη χώρα να τροποποιήσει τον προπολογισμό. Και τελικά, σταδιακά, όλο ένα προς τα εκεί θα σπρώχνουμε. Εγώ νομίζω ότι πρώτα θα πρέπει να δούμε πώς έχει η κατάσταση, να δούμε ποιες προτάσεις έχουμε, πώς θα τις υλοποιήσουμε και κατόπιν να πάμε παραπέρα. Σε ό,τι αφορά το ολοκληρωμένο σχέδιο προϋπολογισμού, έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό, το συζητήσαμε και σήμερα και μάλιστα όταν συζητήσαμε και την έκθεση Γκουλάρ έχουμε τα ευρωμόλογα, το Ταμείο και ορισμένες περιπτώσεις ε, χρειάζονται κάποιες τροποποιήσεις στη συνθήκη και το συζητήσαμε αυτό και στα πλαίσια του ΤΟΥΠΑΚ. Γίνεται λόγος και για τη νομική βάση. Το Συμβούλιο έχει τοποθετηθεί και ο Βαν τοποθετήθηκε με ένα χρονοδιάγραμμα. Πιστεύω ότι στον τριμερή διάλογο για το Τούπακ ίσως εμείς από το Κοινοβούλιο να μην κατορθώσουμε να δώσουμε όθηση, αλλά για την επόμενη σύνοδο θα πρέπει να έχουμε ένα λεπτομερέστερη, μια λεπτομερέστερη εικόνα για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε προς τη λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει λοιπόν καταρχήν να προβλέψουμε κάποιες προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε επί του προπολογισμού και κατόπιν να αποφασίσουμε αν θα δώσουμε τη βοήθεια, αν έχουν γίνει σεβαστές οι προϋποθέσεις. Και τότε να εκταμιεύσουμε τη βοήθεια. Ήθελα την ε, γνώμη σας και γι' αυτό. Κατόπιν, οικονομική ολοκλήρωση. Έχουν γίνει ήδη κάποια βήματα, έχουμε το Europlus, έχουμε και την Ευρώπη 2020, έχουμε το Ευρωπαϊκό Ξάμινο. Ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να βάλουν τη δυνατά τους για να υλοποιήσουν τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για να υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός. Οι συστάσεις που γίνονται και απευθύνονται στα κράτη-μέλη αρκούν έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν στη συνέχεια να προχωρήσουν. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει μια διάκριση μεταξύ των συστάσεων που απευθύνονται στα κράτη-μέλη και τους όρους που τίθενται ή τις συστάσεις που γίνονται, αν θέλετε, για να φτάσουμε σε κάποιες αποφάσεις και να προβλέπουμε κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Σε ό,τι αφορά και πάλι την οικονομική ολοκλήρωση. Τι θα κάνουμε σε ό,τι αφορά ε, τα δημοσιονομικά για την ε, ολοκλήρωση, την δημοσιονομική ολοκλήρωση. πως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε αν θα έπρεπε και η ΕΚΤ ε, να παρέμβει στη φορολογία, παραδείγματος χάρη στη φορολογία των επιχειρήσεων και να κατανοήσουμε πιο συνείς συνέπειες που προκύπτουν σε άλλες χώρες αν εκδηλωθεί πρόβλημα σε μια χώρα και να δούμε επίσης πώς ε, οργανώνεται το σύστημα εποπτείας. Θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά και η Κομισιόν μαζί με το Συμβούλιο θα παρουσιάσει την πρότασή τη και φυσικά και το Κοινοβούλιο θα έχει σχετική έποψη, αλλά είναι σημαντικό να υλοποιηθεί ένα σύστημα που θα εγγυάται πλήρω στο δημοκρατικό έλεγχο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους. και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απόψεις που θα καταθέσετε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε αμέσως, αλλά προηγουμένως θα ήθελα να πω το εξής. Ήδη έχω δει στον τύπο να ονοματίζονται πέντε ευρωβουλευτές που ανέφεραν πράγματα που υποτίθεται ότι είχε πει ο Μάριος Δράγκη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πράγματι τα είπε. Κατά τις διακοπές έγινε αυτό. Και νομίζω ότι είναι θλιβερό γιατί μπορεί ο Ντράγκη να είχε πει το α, το β ή το γ και οι δημοσιογράφοι να ανέφεραν μόνο το β. Αυτό είναι ανακρίβεια λοιπόν. Αλλά αποτελούν ε, πολύ δεν αποτελούν καθόλου έντιμη στάση. Οποιοδήποτε ευρωβουλευτής πήγε και είπε στον τύπο τι δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ ακόμη και αν δεν θεωρούσε ότι ήταν εμπιστευτικό δείχνει έλλειψη σεβασμού για τις διαδικασίες που ισχύουν εδώ μέσα και μπορεί να αποθαρρυνθούν διάφοροι επίσημοι άνθρωποι να ξανάρθουν εδώ να μας μιλήσουν. Και τώρα περνάμε στον εκπρόσωπο των σοσιαλιστών, η Ελίσσα ή ο Λέων Ο Λέων είναι, αλλά θα μιλήσω και εγώ αργότερα αν έχουμε χρόνο. Καλά, ο Λέων ως χιώδης. Ευχαριστώ. Συμμερίζομαι γενικά τις ανησυχίες της Μαριάν Τάισεν ιδιαίτερα ως προς τον δημοκρατικό ή χαρακτήρα διότι το ομοσπονδιακό αυτό άλμα που ζητούν πολλοί δεν πρόκειται να επιτευχθεί αν δεν το δεχτούν και οι λαοί. Ως προς δε τα δημοσιονομικά, οι αντιδράσεις των λαών είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς οι σοσιαλιστές δείξαμε πολύ επικοδομητική στάση στις συζητήσεις για το δίμετρο. Φαίνεται και στα πρακτικά του τριμερούς διαλόγου, αλλά από, τον, από την εξάμετρο από την άλλη μεριά ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε μειωθεί κατά πολύ. Εγώ συμμερίζομαστε λοιπόν και εμείς αυτή την ανησυχία. Ποια είναι η σωστή μέθοδος ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να συνεργαστούν με το, με ευρωπαϊκό για να παίξουν και αυτά κάποιο ρόλο στη διαδικασία. Η λεγόμενη κοινοτική μέθοδος πρέπει να πω ότι παρά το ότι δεν μας βρίσκει για πολύ το σύμφωνος δεν εφαρμόστηκε καν πλήρως. Το θέμα του συναδέλφου Πέτρου Σίμος, Πίτερ Σάιμον, για το τραπεζικό απόρριτο έχει παγώσει στο Συμβούλιο εδώ και ένα χρόνο ενώ το Κοινοβούλιο έχει ήδη αποφαθεί από πολύ καιρό και το Ταμείο Εγγύησης και των Τραπεζών πρέπει κάποτε να συζητηθεί επιτέλους και αυτό. Στην παρουσίασή σας μιλήσατε για κάποιο είδους συντονισμό εξάντε και αυτό μας βρίσκει σύμφωνος από πραγματιστικής απόψεως και αυτό το λέω γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη μακροοικονομική κατάσταση σε αυτή τη συγκυρία να προβλέψουμε περίπου τι μπορεί να γίνει και να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας στην κατάσταση που ισχύει για κάθε χώρα. Η κατάσταση στη Γερμανία δεν είναι ίδια με της Γαλλίας, Ιταλίας ή Ισπανίας. Άρα είναι προφανές ότι εφόσον η συγκυρία, αν η συγκυρία ή όταν η συγκυρία σταθεροποιηθεί, θα δούμε τι θα αποφασιστεί και αν θα εφαρμοστούν όσα αποφασιστούν, τότε θα δούμε αν η ύφεση που αρχίζει σιγά σιγά να εμφανίζεται παντού γιατί τα κράτη-μέλη εδώ και πολλά κράτη-μέλη εδώ και τρεις μήνες γνωρίζουν αρνητική ανάπτυξη όλα αυτά σημαίνουν ότι και οι προτιμήσεις των εκλογέων πρέπει να ληφθούν υπόψη αφού είμαστε δημοκρατικά κράτη. Πρέπει δηλαδή να συνδυάσουμε την αποτελεσματικότητα με τη δικαιοσύνη και με την ίση μεταχείριση. Τώρα για τα δημοσιονομικά ειδικά δεν θα τα πούμε σήμερα όλα, αλλά υπάρχει μια αρχή επί της οποίας εμείς επιμένουμε εκτός από τα ευρωομόλογα που ανέφερε η κυρία Τάισεν και όπου συμφωνούμε επίσης, τουλάχιστον με αυτά που είπε σήμερα, εμείς θεωρούμε ότι η δημοσιονομική δεοντολογία στα κράτη-μέλη πρέπει να συνοδεύεται και με τη θέληση, με κοινοτική επίδειξη θέλησης. Μπορεί να υπάρξει δημοσιονομική ομοσπονδία όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να υπάρχει ομοσπονδιακός προϋπολογισμός. Αν θέλουμε η Τραπεζική Ένωση να υπάρξει και να εφαρμοστεί όπως πρέπει, τότε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να χρηματοδοτηθούν κοινοτικέ πρωτοβουλίες με πολύ πιο μόνιμο τρόπο από ό,τι έγινε για το Σύμφωνο Ανάπτυξης τον περασμένο Ιούνιο. Άρα πρέπει να ξανασυζητήσουμε και το θέμα του κοινοτικού προπολογισμού που δεν ξεπερνάει το 1,2% του κοινοτικού ΑΕΠ αυτή τη στιγμή. Είναι βέβαια επενδυτικό προπολογισμό ή θα έπρεπε να είναι και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διπλασιαστεί και να τριπλασιαστεί και άρα τίθεται και το θέμα των ιδίων πόρων του. Είναι βέβαια, δεν θα το λύσουμε είπα σήμερα, αλλά πρέπει από τώρα να δούμε τι θέλουμε να πούμε. Αυτά προς στιγμή. Πιο συγκεκριμένοι θα γίνουμε σε άλλη φάση. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος από τους ελεύθερους η Σοφία. Ναι, ευχαριστώ Σάρων. Δεν ορίσαμε ακόμη τον εισηγητή μας, αλλά ως συντονίστρια θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα να ξαναπώ στον Επίτροπο αυτά που είπαμε και πριν στον Μισελ Μπαρνιέ και τον κύριο Ντράγκη δηλαδή ότι γνωρίζουμε μεν ότι πρόκειται για πολύ δύσκολα θέματα και πολύπλοκα και η δουλειά μας δεν είναι να σας δυσκολέψουμε τη ζωή αλλά υπάρχει ένα θέμα συνέπειας μεταξύ αυτού που λέμε για τη δημοκρατική νομιμότητα και απ' την άλλη να εγκρίνονται κείμενα χωρίς συναπόφαση. Αυτό είναι λίγο μυστήριο, περίεργο. Ξέρω ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο 127.6 που σας δίνει τέτοια δυνατότητα, αλλά αν είχατε την καλοσύνη να δώσετε και στο Κοινοβούλιο το ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίξει, καλό θα ήταν. Μπορεί να σας έχουμε πιέσει μερικές φορές, αλλά και εμείς σας έχουμε υποστηρίξει ενώπιον του Συμβουλίου. Όπως είπαμε λοιπόν και στους άλλους, δεν θέλουμε θεσμικό πόλεμο ή πόλεμο οργάνων, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να μην γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα και δικαιοδοσίες του Κοινοβουλίου αν συστηματικά η Κομισιόν, ενώ λέει ότι θέλει δημοκρατική μονομιμότητα, παραγωνίζει το Κοινοβούλιο. Όπως ξέρετε, ήμουν εισηγήτρια για το θέμα του συστημικού κινδύνου και ήδη προσπαθήσαμε την κεντρική τράπεζα, στην κεντρική τράπεζα να συνοδευτεί από ένα άλλο όργανο χωρίς να μειώνονται οι δικαιοδοσίες της ούτε η συνέπεια της δράσης της. Μήπως θα μπορούσε η Κομισιόν η Γενική σας Διεύθυνση να μας κάνει μια αντικειμενική αξιολόγηση μετά από δύο χρόνια που υπάρχει το ESRB, τι δούλεψε, τι δεν δούλεψε. Αντί να βιαστούμε δηλαδή να κάνουμε την αναθεώρηση, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ποια είναι η ακριβής αξιολόγηση. Ποιο ρόλο θα παίζει στο εξής. Μακροοικονομικό, μικροοικονομικό. Αν τίποτα δεν το καταλάβαμε καλά να μας το πείτε, αλλά εμείς διαπιστώσαμε ότι Πρόκειται για δομή δυσκίνητη όπου δεν έχει παίξει το ρόλο που θα μπορούσε να έχει παίξει και ότι η ακαμψία αυτή θα έπρεπε να διορθωθεί μέσω μιας καλύτερης επιτήρησης. Σας ευχαριστούμε πάντως για την προσέλευσή σας που τη βλέπουμε ως θέληση συνεργασίας. Ευχαριστώ για τους πρασίνους. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Φανταζόμαι ότι δεν είχατε και πολύ ήσυχο καλοκαίρι. Θα ήθελα να αναφερθώ στα πρώτα σας λόγια. Είπατε ότι θα διαβουλευτείτε μαζί μας. Ε, είμαι παντρεμένος εδώ και 26 χρόνια και νομίζω ότι ένας από τους λόγους ε, που μένω μαζί με τη σύζυγό μου είναι ότι ε, για πολύ σημαντικά ζητήματα δεν είναι ότι διαβουλευόμαστε ένα στον άλλο, αλλά συναποφασίζουμε. Και νομίζω ότι είναι καλή αυτή η συνταγή για ένα γάμο που θα διαρκεί ε, βέβαια, ο καθένα έχει την αυτονομία του, αλλά για τα σημαντικά ζητήματα αποφασίζουμε μαζί. Και θα ήθελα να πω ότι δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι μόνο με τη διαβούλευση. Καθώ ζητείτε την άποψή μα όμω, θα επικεντρωθώ σε θέματα που προσεκτικά έχουν αφαιθεί κατά μέρου και θα προσπαθήσω να ξεκινήσω με κάποιες από τις δηλώσεις σας στην αρχή. Όταν αναφέρατε τη Δημοσιονομική Ένωση, είναι μουσική για τα αυτιά μου όταν μιλήσουμε για δημοσιονομικά θέματα, δηλαδή για τις δαπάνες αλλά και για τα έσοδα και ό,τι έκπληξη το έγγραφο των 5 1 ως Προέδρων είναι σχεδόν αποκλεισ... εντελώς σιωπηρό σε αυτό το θέμα. Ε, και εγώ θα περίμενα η Επιτροπή να πει ότι δεν μπορεί να υπάρχει βιώσιμος προϋπολογισμός χωρίς ε, περαιτέρω και πιο βαθιά δημοσιονομική ολοκλήρωση και στο θέμα της φορολογίας. Θα ήθελα λοιπόν εσείς να τοποθετηθείτε περισσότερο από αυτού και να λάβετε δράση. Δεύτερο σημείο, όταν λέτε ότι πράγματι θα πρέπει να πάμε στην ΟΝΕ δεύτερη έκδοση. Για πολύ καιρό λέμε ότι ε, έχουμε αυστηρούς κανόνες για τον προπολογισμό και το χρέος, αλλά χρειαζόμαστε και αυστηρούς κανόνες και επιθαρκία και για τις επενδύσεις. Και εδώ επισέρχεται η Ευρώπη 2020 και θα περίμενα εδώ τη δική σας ε, Γενική Διεύθυνση για την οδικό σας τομέας να πιέσει τα κρατη για να ε, υλοποιήσουν υποσχέσεις ε, όπως έχουν να κάνουν με τη μείωση της ανέχειας, την παιδεία, τις επενδύσεις, ε, την καταπολέμηση της ανεργίας κτλ. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που λείπει και δημοκρατική λογοδοσία τέλος. Ακούω τι λέτε, ότι πραγματικά έχουμε τώρα αυτό το διάλογο, τον οικονομικό, αλλά δεν μπορεί να αρκέσει, γιατί η Κομισιόν δεν πηγαίνει στα Εθνικά Κοινοβούλια. Εγώ θα έλεγα πολύ ωραίες όλες αυτές τις συζητήσεις. Και φυσικά μου αρέσει να πηγαίνω σε διάφορα μέρη και να συζητώ με του ανθρώπους, αλλά α, αν γνωρίζω ε, ότι μπορεί να συμμετέχω στο παιχνίδι. Βλέπω αλλιώ αυτέ τι συζητήσει. Ε, Παραδείγματο χάρη, κάποιο υπουργό έρχεται εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για μια ωραία συζήτηση, αλλά θα ξέρει ότι δεν θα υπάρχει καμία συνέπεια σε ό,τι αφορά το μέλλον. έχει και ιδιαίτερα κίνητρα να προβεί σε κάποια ισχυρή ανάληψη δράση. Το ίδιο αν πατήσετε στα εθνικά κοινοβούλια, πολύ ωραία, αλλά δεν ε, μπορούν να σας ε, ελέγξουν. Ε, έτσι λοιπόν, η δημοκρατική λογοδοσία ξεκινά με μένα που είμαι υπόλογος ε, στους ψηφοφόρους μου και δεν θα επανέλθω το 2014. Το ίδιο για σας και για τους υπουργούς. Και αυτή παραμένει ε, μια δημοκρατική λογοδοσία ε, μη ισχυρού τύπου. Έτσι λοιπόν, ε, για αυτά που προτείνετε, νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι ακριβώς θεωρείται ως πραγματική δημοκρατική λογοδοσία από το ΕΣΥΑΡ. E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 να τα πω στα αγγλικά. Σκέφτομαι ότι εδώ και 26 χρόνια ο γάμος του Λαμπέρ ήταν πολύ καλό παράδειγμα για τη συναπόφαση που είπε. Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε εύγλωτα για την λεγόμενη δεύτερη Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση που στην ουσία είναι μια τραπεζική ένωση. Και μετά είπατε μερικά γενικότερα ε, τα οποία θέλω και εγώ να σχολιάσω γιατί Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι και εσείς είστε ενήμερος της πιθανής αντίστασης που μπορεί να εμφανιστεί για την Τραπεζική Ένωση. Δηλαδή, η Τραπεζική Ένωση, η πιθανή Τραπεζική Ένωση, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί αν δεν ολοκληρωθεί πρώτα η Δημοσιονομική Ένωση, την οποία επίσης αναφέρατε. Τι σημαίνει όμως αυτό. Ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί θα πρέπει να υποβάλλονται στις Βρυξέλλες οι οποίες θα εξετάζουν τα πάντα και οποιαδήποτε κυβέρνηση δεξιά αριστερή δεν θα μπορεί να προτείνει δομικές αλλαγές χωρίς να υπομείνει την πίεση της Κομισιόν. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να δουλέψει. Αν πρέπει να είναι υποχρεωμένες οι κυβερνήσεις να υποβάλουν τον εθνικό τους προϋπολογισμό στις Βρυξέλλες. Και θα πέσει όλο το φταίξιμο στις Βρυξέλλες ως πηγή του προβλήματος. Δεύτερον, η Δημοσιονομική Ένωση πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια μιας πολιτικής ένωσης. Αυτό θέλω να τονίσω. Η πολιτική ένωση δεν μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς πολίτες. Και είμαι απολύτως βέβαιος γι' αυτό. Όχι σχεδόν βέβαιος και θα υπάρξει μεγάλη αντίσταση όχι μόνο από μερικές κυβερνήσεις αλλά από την τεράστια πλειοψηφία των πολιτών. Ερωτώ λοιπόν απλούστατα. Εσείς κύριε Επίτροπέ μου γνωρίζετε ή συμφωνείτε με αυτό που σας είπα. Και τι μπορεί, τι θα χρειαστεί να κάνει η Κομισιόν για να πείσει τον κόσμο να δεχτεί πλήρη πολιτική ένωση με μία πρωτεύουσα της Βρυξέλλες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλους κοιόδης εδώ. Να περάσουμε λοιπόν στους υπόλοιπους δεν έχουμε πολύ καιρό. Έχω τους κυρίους Μαγκράντη, Περές, Λισαφερέα. Uh, Νομίζω ότι αν μιλήσετε δύο λεπτά ο καθένας θα έχει και ο Επίτροπος πέντε λεπτά για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Κλαουντίο. Συγγνώμη, δεν σε είδα. να επειδή εκπροσωπεί την ομάδα. Παρακαλώ. Πρώτα Μάρτα. Ευχαριστώ. Κύριε Ρέν. Αναγνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη στις ανισορροπίες που αναφέρατε στην ομιλία σας ε, και ε, στο άρθρο σας στη Wall Street Journal η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαράσει τις οικονομικές και νομισματικές πολιτικές την τελευταία δεκαετία και προφανώς αυτοί οι κανονισμοί και οι πολιτικές είχαν αντίκτυπο στην οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω λοιπόν ότι έχετε μια συγκεκριμένη ευθύνη, ένα βαθμό ευθύνης και στο ίδιο άρθρο μιλάτε για αξιοσημείωτη πρόοδο σε αυτές τις ανισορροπίες. Μπορείτε να ορίσετε ποια είναι αυτή η αξιοσημείωτη πρόοδος η Γαλλία σήμερα ε, είπε ότι οι άνεργοι έφτασαν τα 3 εκατομμύρια. Θεωρείτε ότι αυτή είναι αξιοσημείωτη πρόοδος. Και το πρόβλημα μεγεθύνεται και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανεργία. Πιστεύετε ότι η Τραπεζική Ένωση θα επιλύσει το πρόβλημα της ανεργίας? Οι τράπεζες ζητούν διάσωση, αλλά δεν δανείζουν χρήματα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν πιστεύετε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάποια κράτη-μέλη θα τα πήγαιναν καλύτερα εκτός Ευρωζώνης, θα ήταν πιο ανταγωνιστικά και θα μπορούσε η οικονομία τους να μεγεθυνθεί. Σας ευχαριστώ. Να επιστρέψουμε στον Κλάουδιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την ίδια ερώτηση που έθεσα στον κύριο Τράγκη θέλω να θέσω δύο διαφορετικά ερωτήματα για να ε, μας ξεκαθαρίσετε τι γίνεται με τις συνθήκες ε, και πάντοτε αναφέρεστε στο άρθρο 143 το οποίο στην πραγματικότητα μιλά μόνο ε, για την ισοτιμία του ευρώ έναντι των εθνικών μισμάτων, όχι για την δυνατότητα ανάκλησης του ευρώ. Πώς ε, όμως ε, τεχνικά ορίζεται η δυνατό εξόδο από το ευρώ, δηλαδή εγώ θέλω να ρωτήσω είναι δυνατό να βγει κάποιος από το ευρώ ή όχι και διάβασα στην εφημερίδα ότι ο ΣΑ δήλωσε ε, ότι είναι έτοιμο αν η ΕΚΤ αγοράσει τους τίτλους Ισπανία και η Ιταλία καθώς ο, ο ΣΑ ε, τοποθετήθηκε σήμερα κατεπηγόντως είναι σε χειρότερη κατάσταση σήμερα σε σχέση με τα όσα λέγονται στην πραγματικότητα. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, στις ε, παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε μακροπρόθεσμα, με όραμα, σχεδιασμό, χρονοδιάγραμμα για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη και βραχυπρόθεσμα. Και πιστεύω ότι τα βραχυπρόθεσμα είναι επίγοντα. Βλέπουμε ότι η κρίση της Ευρωζώνης έχει χτυπήσει και την καρδιά της Ευρωζώνης. Μπορεί να πλήττονται ιδιαίτερα οι χώρες του Νότου, αλλά ήδη στη Γερμανία μειώνονται οι εξαγωγές, ε, ε, Ήδη βλέπουμε ότι έχει επιπτώσει τη βιομηχανική παραγωγή, στην αγορά εργασίας. Η Γαλλία έχει άσχημη κατάσταση επίσης, το είπε συνάδελφό μα, στην αγορά εργασίας και στη βιομηχανική της βάση. Ήθελα να σα ρωτήσω, η, η κατάσταση στην Ισπανία και στην Ιταλία, η, πιθανότητα προσφυγής στο μηχανισμό, έχει κοστολογηθεί, έχει, έχετε εναλλακτικά σενάρια, πώς θα επιδράσει στην κατάσταση αυτή. Και τα έχετε υπόψη σχεδιάζετε παράλληλα μέτρα με τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής που θα δίνανε αναπτυξιακές επνοές. Ο, ο Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ολλανδίας ανέφερε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να πάρει προκαταβολή από την αναμενόμενη δόση του δανείου για να μπορέσει να θέσει σε εφαρμογή κάποια σχέδια αναπτυξιακά πέρα από την αναμενόμενη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Ε, αντιμετωπίζετε τέτοια τέτοια θέματα, προγράμματα άμεσης παρέμβασης λόγω της επιδεινόμενης κατάστασης σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ευχαριστώ, Περβάνης. Ευχαριστώ, κύριε πίτροπε. Ξέρω ότι το χαρτοφυλάκιό σα, ε, μάλλον ε, σας οδηγεί στο να κάνετε αυτές τις ε, προτάσεις ενώπιον μα, όμω ανήκετε και σε ένα σώμα που θα πρέπει να συμβάλλει ή να αντιδράσει απέναντι στο πεδίο που καλύπτει η έκθεση της συναδέλφου Τίσεν λαμβάνοντα υπόψη και την πρόταση του Περοπόη το Δεκέμβριο. Όμω, μένα με εκπλήσουν δύο πράγματα. Καταρχήν, κατανοώ ότι στην ομάδα του Βάρουν Πόη αυτό το θέμα συνεχίζει να θεωρείται ότι πρέπει να είναι οικονομολόγοι αυτοί που το διαχειρίζονται. Η δική μου αντίληψη είναι ότι αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε θα συνεχίσουμε να έχουμε μέτρα, ιδιαίτερα προκυκλικά, όπως είχαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Και όταν ε, λέω ιδιαίτερα προκυκλικά μέτρα, δηλαδή μιλάμε για τα μέτρα λιτότητας ε, που ουσιαστικά μας οδηγούν σε επιδείνωση της κατάστασης. Ας ε, υπαναχωρήσουμε λίγο για να δούμε ποιο είναι το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε. Μία κρίση που γεννήθηκε στις ΗΠΑ και μας καταβροχθίζει, μας καταπίνει. Και για να χρησιμοποιήσω ένα πιο γεωγραφικό όρο, αλλά που νομίζω ότι είναι μια ισχυρή εικόνα, έχω την εντύπωση ότι ε, ουσιαστικά ε, βρισκόμαστε σε μία ε, ρόδα που γυρίζει συνεχώς και θα, για να βγούμε από αυτή τη ρόδα που γυρίζει συνεχώς θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο ορίζοντα και αυτός είναι ο χάρτης πορείας που θα πρέπει να κατατεθεί το Δεκέμβριο γιατί διαφορετικά ε, όλα τα συστατικά που επέτρεψαν στους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που επέτρεψαν ε, στην γενιά που προηγήθηκε της δικής μου. Να εφεύρουν, να φανταστούν ε, και να ελοποιήσουν ε, την ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, όλα αυτά θα διαλυθούν. Και όταν έρχεστε εδώ να μας πείτε Α, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο έλεγχος Συγγνώμη, δεν θέλω να σας μιμηθώ έτσι, δεν μιλάτε έτσι περαιτέρω έλεγχη, περαιτέρω ε, δημοσιονομική νοπιστή και θα μιλήσω στα οικονομικά κοινοβούλια και θα του εξηγήσω ότι αν αποκλίνω από του προπολογισμού, τότε αυτό δεν αρκεί, τότε αυτά δεν θα λειτουργήσουν. Γιατί έτσι θα ευνοηθεί ο ρατσισμός, η ξενοφοβία ε, και η εχθρότητα μεταξύ των κρατών. Ξέρω ότι έχουμε μια θεμελιώδη συζήτηση, αλλά αν ε, πρέπει να διακόψω, θα διακόψω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πίτροπε. Εγώ είχα πολλές ερωτήσεις να σας θέσω, αλλά θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Μία πρώτη ερώτηση. Όταν μιλάτε για μία νέα ονέ, εγώ χαιρετίζω ε, αυτή τη σκέψη. Είναι ιδιαίτερα απαραίτητη αυτή η νέα Οικονομική και Νομισματική Ένωση, αλλά δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ισχυρή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν, στο νομοθετικό πλαίσιο όπου θα γίνουν όλες αυτές οι τροπήσει, θα πρέπει να εκπροσωπούνται και οι πολίτες. Δεύτερο σημείο σε σχέση με τον έλεγχο του δημοσίου χρέους. Το Κοινοβούλιο έλαβε διάφορες αποφάσεις για το θέμα αυτό. Και εγώ νομίζω ότι ο κύριος Επιτρόπος επίσης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να υπάρχει κοινή έκδοση ομολόγων. Όμως κάτι που δεν κατάλαβα εγώ καλά είναι με ποιο τρόπο είναι στις παρεμβάσεις ε, που προβλέπονται για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι διαρθρωμένες με, πώς διαρθρώνονται με αυτό το ευρύτερο πλαίσιο της έκδοσης ε, κοινών ομολόγων. Δηλαδή γίνεται ένας υπολογισμό βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, αλλά όλα αυτά δεν είναι ξεκάθαρα. Εγώ θα ήθελα να μας τα αποσαφηνίσετε αυτά. Κατόπιν, τρίτο σχόλιο για τον δημοσιονομικό έλεγχο, για τη Δημοσιονομική Ένωση. Πιστεύω ότι δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει χωρίς να αγγίξει το θέμα των φόρων, των φορολογικών εσόδων. Και επίσης ε, δεν πιστεύω ότι είναι δυνατό να επιτρέψουμε μέσα σε μια νέα αγορά να συνεχίσουν να υπάρχουν ε, πολλές ε, τέτοιες συμπεριφορές κοινωνικού φορολογικού ντάμπινγκ. Εμείς θα πρέπει να δημιουργήσουμε ίσους κανόνες για όλους ε, και για τη φορολογία και για τα κοινωνικά ζητήματα και να ξαναδούμε πώς θα ευνοήσουμε τον ανταγωνισμό. Ξέρω ότι δεν έχω χρόνο. Ήθελα 10 δευτερόλεπτα μόνο για να θέσω μια ερώτηση ακόμη στη χώρα μου, στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία ακολουθεί τις συστάσεις της Κομισιόν ε, της Τρόικας. Πολύ στενά και δεν λειτουργούν τα πράγματα. Το μόνο που λειτουργήσε ήταν η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Γιατί, ξέρετε, με την ύφεση δεν υπάρχουν εισαγωγές, και βελτιώνεται το εμπορικό συζύγιο. Έχουμε 16% ενεργεία, 30% στους νέους και έχουμε ύφεση που είναι εγκατεστημένη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δέχεται, θα δεχτεί να αναθεωρήσει αυτή τη συνταγή που χρησιμοποιεί τώρα ή θεωρεί ότι ανεξάρτητα αποτελέσματα είναι μία και μόνη συνταγή. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Δεν κατάλαβα γιατί οι σοσιαλιστέ πάντα δεν περιορίζονται στα δύο λεπτά. Για να δούμε η Άννη μήπω θα καταφέρει καλύτερα. I will, I've done much in the previous... Θα τα καταφέρω, γιατί έχω κάνει πολύ περισσότερα στην προηγούμενη συζήτηση. Πρώτο μέρος της ερώτησης, η Επίτροπε, πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση όπως η ερώτηση της Ελίζας. Μιλάμε για ποιοτικά μέτρα για την ε, Δημοσιονομική Ένωση. Στην τωρινή πρόταση όμως ε, έχουμε ποιοτικά μέτρα που κινούνται στα ανώτατα όρια και στα... Ε, ε και, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για πολιτικό συντονισμό σε κέρυες πολιτικές όπως το φορολογικό σύστημα, τα κοινωνικά συστήματα και αναρωτιέμαι αν προτίθεστε να συμπληρώσετε την τωρινή πρόταση για το πλαίσιο του προϋπολογισμού με προτάσεις που θα αφορούν φορολογία και κοινωνικά συστήματα. Επίσης, κύριε Επίτροπε, ενημερώστε μας λίγο σε σχέση με τη συνέχεια που δόθηκε στις αποφάσεις για την, της ε, κορυφής για την άμεση η απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον ESM, το μηχανισμό για να σπάσουμε το φαύλο κύκλο, όπως είπατε, μεταξύ, ε, στις σχέσεις μεταξύ ε, κυβερνήσεων και τραπεζών. Και το ερώτημα είναι, όταν ας πούμε βάλουμε τους όρους σχετικά με το ποιες θα είναι οι επιλέξιμες τράπεζες για να συμμετέχουν σε αυτή την ανακεφαλαιοποίηση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την αποτελεσματικότητα των, ροπεζών, των κυβερνήσεων. Γιατί ε, υπάρχει ο κίνδυνος να μην σπάσει ο φαύλος κύκλος, αλλά να ενισχυθεί ο φαύλος κύκλος μεταξύ τραπεζών και ε, κυβερνήσεων. Και θα υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά και δύο ε, ε, ομάδες τραπεζών μέσα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες και τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, ο τελευταίο που είχε ζητήσει το λόγο δεν βρίσκεται εδώ, οπότε δίνουμε κατευθείαν το λόγο στον Επίτροπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχήν, ε, σας ευχαριστώ πολύ για την ουσιαστική συζήτηση που είχαμε σήμερα και για τις απόψεις που καταθέσατε. Είχαμε πολύ μεγάλη συνεισφορά από την πλευρά σας για την περαιτέρω προετοιμασία των προτάσεων αυτών. Και βλέπω ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση πολύ σύντομα για την ε, νέα οικοδόμηση της ΟΝΕ και για την οικοδόμηση μιας ε, τραπεζικής ένωσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις στα 4,5 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου. Έτσι λοιπόν θα επικεντρωθώ στο σημερινό θέμα. Θα θυμάστε ότι η σημερινή συζήτηση εδώ αφιερώθηκε στο πώς θα προχωρήσουμε προς μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση και θέλω να υπενθυμίσω ότι θα υθετήσουμε την νομοθετική μας πρόταση για την Τραπεζική Ένωση σε 10 ημέρες περίπου. Έτσι λοιπόν, συνεχίζονται οι στην Κομισιόν. Το καλοκαίρι εργαστήκαμε πάρα πολύ εντατικά και συνεργαστήκαμε στενά και φυσικά με τον πρόεδρο Περόσο και με το φίλο και συνάδελφο Μισελ Μπαρνιέ και πολλού άλλου συναδέλφου και το Χακίν Ελμούνια. Και οι υπαλληλοί μα τι δύο τελευταίε εβδομάδε εργάστηκαν βάση πολιτικής καθοδήγησης που δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο, προκειμένου να έχουμε μια έγκαιρη και ουσιαστική υιοθέτηση της πρότασης για την Τραπεζική Ένωση για να μπορέσουμε να σας την παρουσιάσουμε σε δύο εβδομάδες και να μπορούν να ληφθούν οι αποφάσεις μέχρι τα τέλη του έτους. Το πρώτο σημείο, το πρώτο σχόλιο που έθεσε η εισηγήτρια αλλά και άλλοι συναδέλφοι για την νομική βάση. Κατανοώ τις ανησυχίες σας ε, σχετικά με το θέμα αυτό. Σκοπεύουμε να καταθέσουμε τις ακόλουθες ε, νομοθετικές προτάσεις στο πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου. Μία πρόταση κανονισμού για τη σύστοση του ενιαίου αποπτικού μηχανισμού που θα βασίζεται στο άρθρο 127.6 και κατόπιν μια πρόταση που θα βασίζεται στο άρθρο 114 που θα τροποποιεί τον κανονισμό EBA της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για να διασφαλίσουμε πραγματική λεπιδράση μεταξύ της EBA της ε, νέας εποπτικής αρχής και των κρατών μελών που δεν συμμετέχουν ακόμη στην Τραπεζική Ένωση και για να έχουμε διατάξεις που θα μπορούν ε, να εφαρμοστούν για τις εξουσίες, της αρμοδιότητες ε, του μηχανισμού εποπτείας. Παράλληλα, θα θετήσουμε μία ανακοίνωση που θα παρουσιάζει την άποψη της Κομισιόν για την Τραπεζική Ένωση συνολικά, στο σύνολό τη, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων ε, για την κατάθεση των εγγύσεων και για την εξυγίανση των τραπεζών. Θα έχουμε λοιπόν και ένα μηχανισμό για τη διάσωση, ένα ταμείο διάσωση των τραπεζών και το σύστημα διασφάλισης των καταθέσεων. Αυτό είναι ένα σχέδιο και να υπογραμμίσω ότι στο πλαίσιο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει ισχυρή φωνή επί του αποτελέσματος και θα θυμάστε ότι πριν να μπορέσουμε να εξετάσουμε νέα βήματα προς ε, το δεύτερο στάδιο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε πράγματι να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο μηχανισμό αποπτίας. Και αυτό σχετίζεται με τα σχόλια που ακούστηκαν από πολλά μέλη του Κοινοβουλίου, την κυρία Φεραίρα, την κυρία Ποδηματά, την κυρία Γκουλάρ, τον κύριο Λαμπερτ σε σχέση με τη συσχέτιση με την ε, άμεση ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Καταρχήν, χρειαζόμαστε τον νέο αποπτικό μηχανισμό που πρέπει να τη σε ισχύ, πρέπει να καταστεί επιχειρησιακός, και κατόπιν ε, θα έχουμε την άμεση επαγγελματιοποίηση των τραπεζών. Φυσικά δυνάμει μιας ε, κανονιστικής απόφασης που θα ληφθεί σύμφωνα με τους κανόνες του SSFF. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να κινηθούμε αποτελεσματικά και γρήγορα και προς αυτό εργαστήκαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά, να συνεργαζόμαστε εντατικά με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προκειμένου να έχουμε μια εγκαιριοθέτηση της πρότασης αυτής. Να προσθέσω ότι βάσει εμπειρία δύο σημαντικών νομοθετημάτων, το πακέτο για πιο ισχυρούς ε, κανόνες ε, εποπτείας ε, και πρόληψης και το Six Pack για ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση. Νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ευγνώμονες στο Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της νομοθεσίας που προτείνεται. Έτσι λοιπόν, καλωσορίζω μια ισχυρή συμβολή και συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μελλοντική πρόταση για την Τραπεζική Ένωση και τη συζήτηση αυτού του πολύ σημαντικού νομοθετήματος. Σε ό,τι αφορά άλλα θέματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Σχετικά με τον ακριβή σχεδιασμό της ΕΚΤ, του ενιαίου προληπτικού μηχανισμού της ΕΚΤ. Εκεί υπήρξαν και κάποιες ερωτήσεις, όπως ε, η συμμετρία των καταθέσεων και της εξυγίανσης με την εποπτεία και πώς θα διασφαλίσουμε τη λογοδοσία στην εποπτεία ενώ θα διατηρήσουμε την ανεξαρτησία στην ε, νομισματική πολιτική. Αυτά είναι σημαντικά θέματα και θα πρέπει να επανέλθουμε. Έχουμε εσωτερικέ ε, συζητήσει επί του παρόντο για τα θέματα αυτά. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ενοποιημένο σύστημα που θα έχουμε και τον ε, μηχανισμό εποπτείας και τα στοιχεία του δεύτερου σταδίου, δηλαδή το σύστημα αγγίσης καταθέσεων και το Ταμείο Εξηγένσης των Τραπεζών για τις τράπεζες και τα κράτη-μέλη. Και εδώ συμφωνώ μαζί σας ότι δεν θα πρέπει να αφορά μόνο την Ευρωζώνη αυτό, αλλά και τα κρατη που δεν αποτελούν ακόμη μέρος της Ευρωζώνης, αν δεσμευτούν νομικά, και είναι έτοιμα να συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα, σε αυτή τη βάση, τότε θα πρέπει να είναι ανοιχτό αυτό το σύστημα και για εκείνα τα κράτη-μέλη. Μπορεί παραδείγματο χάρη να σκεφτείτε την περιοχή της Βαλτικής ε, της Σκανδιναβία. Υπάρχει ένα σχεδόν ε, ολοκληρωμένο ε, σύστημα τροπεζικού τομέα. Υπάρχουν χώρες της Ευρωζώνης όπως η Φιλανδία, η Εστονία, ε, αλλά έχουμε και άλλες χώρες, ε, Λετωνία, Λιθουανία, που δεν έχουν πει ακόμη και έχουμε και μια χώρα, τη Σουηδία, που έχει απορρίψει την ε, συμμετοχή στην Ευρωζώνη με δημοψήφισμα και έχουμε και τη Δανία, που δεν ανήκει στο ευρώ. Και έτσι λοιπόν θα είχε νόημα να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε εμπόδια που δεν είναι απαραίτητα σε οποιαδήποτε μέρος της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα αποτελεσματικό μηχανισμό βοηθείας για τις τράπεζες της Ευρωζώνης. Πολλές ερωτήσεις θα πρέπει να απαντηθούν σε μελλοντικέ ε, συναντήσεις. Ευχαρίστως να επανέλθω και να συζητήσω μαζί σας και εδώ στην Ολομέλεια. Τα θέματα που τέθηκαν ε, από συναδέλφους που αφορούν την ανάπτυξη είναι ζωτικά. Και μην υποτιμάτε τη σημασία των αποφάσεων που, λαμβάν, που ελήφθησαν στο τελευταίο Συμβούλιο του Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά το χάρη το πώς θα προχωρήσουμε για να αυξήσουμε το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να προωθήσουμε τις ε, δημόσιες επενδύσεις στην Ευρώπη, ε, για τις υποδομές, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές και επίσης ε, να δώσουμε και κίνητρα για να υπάρξουν ιδιωτικές επενδύσεις, γιατί αυτό χρειαζόμαστε προκειμένου να ξαναρχίσει η ανάπτυξη στην Ευρώπη και να επανέλθουμε στην βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασία στην Επιρώμας. μας. Θα ήθελα να κλείσω εδώ και όπως είπα θα επανέλθω σύντομα για να συνεχίσουμε αυτή την πάρα πολύ σημαντική συζήτηση για το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, αλλά και για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι βέβαια ότι θα γίνουν και πολλές άλλες συζητήσεις, όπως είπατε, και επίσημα και άτυπα το χρονοδιάγραμμα προς το παρόν είναι να εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης στις 19-20 Σεπτεμβρίου με προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 24 Σεπτεμβρίου για να συζητηθούν στις 8 οι τροπολογίες και 15 Οκτωβρίου να ψηφιστεί και να πάει τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια. Πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα, αλλά πρέπει να κινηθούμε ταχύτατα. Ευχαριστώ που το δεχτήκατε αυτό το τόσο ε, δύσκολο χρονοδιάγραμμα και τη Μάριαν. Και δίνω πάλι την Προεδρία στον Πάμπλο. Por favor, continuamos. Συνεχίζουμε με το σημείο 11. Παρουσίαση του σχεδίου έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και καθώς έχουμε ξεφύγει εντελώ από το πρόγραμμά μας, να δώσουμε κατευθείαν το λόγο στον κύριο Γκοζές που είναι ο εισηγητής. Έχει το λόγο, Ζανπόλ. Monsieur le Président, je vous remercie. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα θα μιλήσουμε πράγματι και κλεισμένων των θυρών γιατί δεν θα μας ακούσει κανείς. Άρα δεν θα υπάρχουν και διαρροές. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος. Και για μας και για τους ε, διερμηνείς που δουλεύουν από τις 2.30. Το πρόγραμμα το έχετε να σας πω το γενικότερο πλαίσιο, η οικονομική και κοινωνική κρίση και η χρήση του χρέους και η κίνδυνη να επεκταθεί από τη μία χώρα στην άλλη. Αυτό μας όθησε να δημιουργήσουμε τη διαδικασία αυτή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που τώρα θα επαναλάβουμε. Λοιπόν, η έκθεση λαμβάνει υπόψη της τις συζητήσεις που έκανα με τους διάφορους σκιώδεις και τις προτάσεις τους. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο επιτρέπει προηγούμενη συνεννόηση στην Ευρωζώνη για να μειωθούν οι κίνδυνοι επέκτασης της κρίσης Τα μέτρα έχουν πάντα σαν στόχο τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών μέτρων, την προώθηση της ανάπτυξης και τονίζουμε ιδιαιτέρως ότι οι συστάσεις αυτές δεν είναι καθολικές αλλά πολύ συγκεκριμένες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων. Για να μην μπορεί ένας αρχηγός κράτους να πει ότι έκανε ό,τι έπρεπε χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Προσπαθήσαμε να δούμε ποιες δομικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη. Ζητούμε από την Κομισιόν να παρακολουθήσει στενά την εφαρμογή τους και να κάνει αξιολογήσεις που να είναι χρήσιμες και για την επόμενη περίοδο και προτείνω να ζητήσουμε από τις χώρες μέλη να τηρήσουν αυστηρά τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητα όπως τροποποιήθηκε από την εξάμετρο. Θα έπρεπε σύντομα να συμφωνήσουμε και για την δίμετρο και μετά θα αρχίσει καινούργιο τριμερής διάλογος για τα δύο κείμενα της Ελίζα Φερέρα και του δικού μου. Αυτά είχα να σας πω σήμερα προκαταρκτικά, τώρα θα ακούσω τι έχετε να μου πείτε εσείς. Αλλά υπενθυμίζω ότι ήδη έχω αναφέρει πολλές από τις ιδέες σας, με την άδειά σας βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκοζές. Η κυρία Φερέιρα, εξ ονόματος Σοσιαλιστών, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω ένθερμα τον κύριο Κουζές για το πόσο τακτικά συνέταξε το κείμενο στα πλαίσια συνεχούς διαλόγου με τους κοιόδης εισηγητές. Και επίσης θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί ήταν επικοδομητικός ο διάλογος αυτός, δηλαδή όχι απλώς μας άκουσε, αλλά πολλές από τις προτάσεις ε, και τα θέματα που σας το κοινού τα συμπεριέλαβα στην έκθεσή σας. Ευχαριστούμε λοιπόν για την επικοδομητική μέθοδο που χρησιμοποίησατε για να συντάξετε το κείμενο. Φυσικά εγώ ταυτίζομαι πολύ περισσότερο με αυτή την πρόταση κειμένου σε σχέση με την αρχική, για λόγους που ήδη έχω επισημάνει. Φυσικά διατηρούνται κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις ε, μεταξύ των διαφοροποιήσεων. Μιλώ για κάποιες αποχρώσεις Ίσως δεν θα ήμουν τόσο ενθουσιώδης εγώ στις παραγράφους 3, 9 και 10, αλλά αυτές ε, είναι και διαφορές πολιτικής φύσεως. Αν θέλουμε να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό δεν είναι τόσο σημαντικό. Ίσως ε, αν ήταν ε, δυνατό να κάναμε μία αναφορά σε σχέση με τις συστάσεις που γίνονται στις χώρες πιο επίμονα για να υπάρχει πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Γιατί αυτός ο παράγοντας είναι πάρα πολύ σημαντικός για να μην υπάρχουν ε, κοινωνικές αδικίες. Κυρίως όταν λαμβάνονται μέτρα μεταρρύθμισης, μεταρρυθμιστικά μέτρα, όπως ε, είναι αυτά που συζητούνται και λαμβάνουν χώρα σε πολλές από τις χώρες μας. Ένα ακόμη σχόλιο. Σχετικά με την αναγκαιότητα να προσεγγίσουμε την Ευρωζώνη ως σύνολο και επομένως ε, να γίνονται κάποιες συστάσεις όχι μόνο στις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και που πρέπει να προσαρμόσουν την οικονομία τους, αλλά να επιτρέπεται να δίνεται και κάποια κίνητρα στις άλλες χώρες ε, να βοηθήσουν ε, τους ε, άλλους να δίνουν ε, ουσιαστικά οξυγόνο στις άλλες χώρες. Αυτή είναι μια συνέπεια της ανάλυσης που κάναμε από κοινού στο πλαίσιο του Sixpack. Και τέλος, αναγκαιότητες, συστάσεις που γίνονται είτε την είτε στην περίπτωση ε, της ε, Τρόικας, ε, που γίνονται από την Τρόικα δηλαδή, να μην θεωρούνται ως μια δικτατορική επιταγή ή να διατηρούνται άφικτες για πάντα, αλλά να υπάρξει και μια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. Εγώ μιλώ για κανόνες που προτείνονται σε μια χώρα, αν ε, μια μεγάλη χώρα εταίρος ε, μπει σε ύφωση, ε, φυσικά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το μέγεθος της χώρας. Έτσι λοιπόν, εγώ θα ήθελα η ανάλυση αυτή να είναι πιο λεπτομερής όπως είπε και ο κύριος Γκοζές, αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα και να μην θεωρείται ως κάτι που θα παραμείνει στο δυναικές, αλλά να μπορούν να γίνουν κάποιες προσαρμογές και διορθώσεις ανάλογα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Αυτές είναι ορισμένε από τις προτάσεις. Το κείμενο θεωρώ ότι βελτιώθηκε σημαντικά και ευχαριστώ τον κύριο Γκοζές για το έργο του. Και Ελπίζω να διατηρηθεί αυτό το θετικό πνεύμα συνεργασίας μέχρι την τελική έγκριση της έκθεσης και θα καταθέσω και κάποιες τροπολογίες από τη δική μας πλευρά προς την κατεύθυνση που μόλις σας εξέθεσα. Ευχαριστώ πολύ από τους φιλελευθέρους. Η κυρία Γκουλάρ. Euh. Ευχαριστώ τον Ζαν Πολ για όσα έκανε. Θα είμαι σύντομη γιατί είναι αργά και όλο το απόγευμα λέγαμε πώς να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση αλλά τελικά σαν το σύσυφο πάντα την ίδια πέτρα προσπαθούμε να σμπρώξουμε λοιπόν και μας ξαναπέφτει κάτω για να συνδέσουμε τα πράγματα με την έκθεση της Μαριάννας πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια υπάρχει βέβαια και το δίμετρο Συμφωνώ με αυτά που είπε και η Ελίζα προηγουμένως. Όλο το θέμα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής είναι σημαντικό. Και είπαμε οι βελτιώσεις να μην βλάπτουν τελικά τον προϋπολογισμό. Αλλά να τα δούμε τα πράγματα πιο λεπτομερώς. Ευχαριστώ Ζαμπόλ και θα συνεχίσουμε τις συνεννοήσεις. Ευχαριστώ Σιλβί. Από το ECR νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς. Έτσι λοιπόν να δώσουμε το λόγο στην κυρία Τουρούνεν που εκπροσωπεί τους πράσινους. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. και για τη χρονική στιγμή που είναι ωραία μετά τις διακοπές. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Η πράσινη είναι πολύ υπέρ της ιδέας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, διότι οδηγεί σε ισχυρότερη, υγιέστερη οικονομική διακυβέρνηση στην Ένωση. Αλλά χρειάζονται και κάποιες διορθώσεις και υπάρχουν και μερικές ανισορροπίες που πρέπει να τις ε, αποκαταστήσουμε γιατί δεν έχουν αποκατασταθεί. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη απαριθμώντας τις. Πρώτον, δεν ζητάμε ή δεν θα έπρεπε να ζητάμε από τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν αυστηρή πειθαρχία μόνο σε ό,τι αφορά τις δημόσιες δαπάνες, αλλά θα πρέπει να ζητούμε από τα κράτη-μέλη να έχουν και μια ε, σωστή εξυγίανση, όχι κυκλική, προκυκλική. Και αυτό γίνεται τώρα. Θα πρέπει να διορθωθεί η Ευρωζώνη, η Ευρώπη των 27. Αυτό δεν μπορεί να γίνει βραχυπρόθεσμα, δεν θα ήταν έξυπνο αυτό, ούτε αντικατοπτρίζει θα αντικατόπτριζε την οικονομική πραγματικότητα σε κάθε χώρα. Όχι χρειάζεται όχι μόνο αυστηρότητα, αλλά και εξυπνάδα και ευελιξία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Δεύτερον, βλέπουμε ότι κάποιες συστάσεις ή ότι οι συστάσεις μάλλον δεν ε, ισορροπούν σε σχέση με τις ε, χαμηλότερες συντάξεις, ε, το πρόβλημα των κοινωνικών δαπανών, επίσης άλλα θέματα, ε, ε, κέρδη από κεφάλαια, κεφαλαϊκά κέρδη, ε, που δεν λαμβάνονται ισομερώς υπόψη στις, ή το φορολογικό, δεν λαμβάνεται υπόψη. Τέλος, θα έπρεπε να διατηρηθεί η διαφορά μεταξύ στόχων και μέτρων. Υπήρχε και στην έκθεση Μπερές η διάκριση αυτή και στην πρώτη σας έκθεση, ούτω ώστε να υπάρχει μια πολιτική ευχέρεια, μια ευχέρεια πολιτικής, ε, ενώ ε, καλύπτεται η πολιτική τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Για να τελειώσουμε, δεν υπάρχει κανείς από την ΚΟΕ. Να περάσουμε λοιπόν στον κατάλογο των ομιλητών. Μόνο ο κύριος Λούντβικσον έχει ε, ζητήσει το λόγο. Αν θέλει κάποιο άλλο το λόγο, τώρα παρακαλώ να το ζητήσει ο κύριος Λούντβικσον. Ευχαριστώ. Πρέπει να καταδείξουμε τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο βελτιώνεται, λειτουργεί όλο και καλύτερα, αλλά πρέπει να λυθούν και κάποια προβλήματα εδώ. Και κάποια μέτρα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα. Ένα πρόβλημα είναι ότι η Κομισιόν στις συστάσεις που κάνει σε κάθε χώρα ε, ναι, τίνει να επισέρχεται στην αγορά εργασίας και στην αυτονομία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων. Λοιπόν, ε, ξανά και ξανά καλεί τα κράτη-μέλη να ε, μειώσουν τους μισθούς. Ε, δεν είναι αποδεκτό αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια αυτονομία στις συλλογικές διαπραγματεύσεις που πρέπει να γίνει σεβαστή για να λειτουργεί και η αγορά. Κάθε επίθεση σε αυτή την αυτονομία αντιφάσκει σε βασικά συνδικαλιστικά δικαιώματα. Και υπάρχει αυτό, το ξέρει και η Κομισιόν το, και υπάρχουν και ε, τα νομικά μας κείμενα και στο Κοινοβούλιο ε, υπερασπιζόμαστε εμείς αυτήν την ε, συνδικαλιστική αυτονομία και στα πλαίσια του δέσμη των 6 και της δέσμη των 2 μέτρων. Η Κομισιόν πρέπει να αλλάξει τη θέση της εδώ. Επίσης, ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα πρέπει να επικεντρωθεί στη φοροδιαφυγή και αποφυγή με μέτρα αποτελεσματικά γιατί με τα χρήματα από τη φοροδιαφυγή μπορούμε να βοηθήσουμε να καταπολεμηθεί η κρίση. Πολλές φορές χάνονται πάρα πολλά ποσά. Ε, ενίσχυση λοιπόν της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Αυτό πρέπει να είναι πολύ κεντρικό θέμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο πολύ σύντομα και στα γερμανικά για τον Ζαν Πολ και για τους άλλους γερμανόφωνους. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Ευχαριστώ που τονίζετε ένα θέμα ιδιαίτερα, δηλαδή ότι μόνο εν μέρη έχουν τηρηθεί οι μεταρρυθμίσεις που υποσχέθηκαν τα κράτη-μέλη. Ο κατάλογος είναι μακρός και δημιουργεί πρόβλημα. Είναι πολλέ οι μεταρρυθμίσει που δεν έγιναν και από πίσω κατά κανόνα κρύβονται κράτη που ποτέ ε, δεν δεν προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ε, Ε, υπάρχουν όμως και χώρες ε, που βρίσκονται λίγο κάτω από το όριο και δεν, ε, πιάνουν, δεν αναφέρονται από την Κομισιόν. Καλό θα ήταν λοιπόν να κρατήσουμε μια ενιαία στάση απέναντι στις χώρες. Υπάρχει και ένας άλλος τομέας που πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις. Δηλαδή το ευρωπαϊκό εξάμεινο που πρέπει να συνδεθεί στη στρατηγική Ευρώπη 2020 ε, βάζοντας την έμφαση στην ε, βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση αλλά και τους άλλους στόχους της Ευρώπης 2020 πρέπει να τους εντάξουμε στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και μετά στο ευρωπαϊκό εξάμεινο θα αξιολογούνται. Και εδώ υπάρχουν ανισότητες και νομίζω ότι ε, είναι σημαντικό να το ε, τονίσουμε αυτό. Υπάρχει και κίνδυνος ε, κάποιες σημαντικές, κάποιες σημαντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις να χαθούν, όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Φτώχειας, που μέχρι τώρα συνεργάστηκε πολύ και ήλπιζε να κερδίσει από αυτή τη στρατηγική. Αλλά τώρα δυσανασχετεί γιατί δεν περιλαμβάνονται προτάσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας, οπότε τι, δεν βλέπει νόημα να συνεργάζεται. Ε, αλήθεια, σωστό είναι αυτό. Άρα είναι σημαντικό εμείς ως Κοινοβούλιο να φροντίσουμε να είναι ε, ισότιμα τα μέτρα ε, ε, και ισότιμα τα μέτρα για την αντιμετώπιση κάθε στόχου. Ευχαριστώ για να ολοκληρώσουμε. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Την επόμενη φορά λέει ο Πρόεδρος. Για να ολοκληρώσουμε. Ο εισηγητής ε, έχει το λόγο. Παρακαλώ, Ζανπόλ. Ευχαριστώ. Λίγες παρατηρήσεις θα κάνω. Θα διαβάσω τις ε, τροπολογίες ε, και θα τις εντάξω στο έγγραφο. πάντοτε, πάντοτε είμαι πρόθυμος να συμμετέχω σε ε, καλές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ και καλό σας βράδυ. Perdón. Σας ευχαριστώ όλους. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ε, είναι η 11η Σεπτεμβρίου. Η συζήτηση θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 8 Οκτωβρίου και στην Ολομέλεια 22 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε αύριο. Thanks to you.